Bene. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας ε, αναμεταδίδεται μέσω του ίντερνετ και ξεκινώ με τον ορισμό των εισηγητών για αποφάσεις σχετικές με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Έγινε η πρόταση χτες στην ε, συνάντηση των συντονιστών, η αντιπροσωπεία στην Ιταλία για το ΕΛΚΑ, Μέντελς Ντεβίσκο, Σαλάτο και ε, εγώ πρόεδρος για τους σοσιαλιστές Ερέρο, Μάρτιν και Κουαρτιέρη, εκτός ποσοστώσεων γιατί είναι Ιταλός και ε, μέχρι τον κύριο Μέσερ Σμιτ για την Κοπενχάγη εκτός από μένα από δύο βουλευτές από το ΕΛΚΑ και δύο από τους Ελιστές έναν Άλντε και από τον Σόντεργατ και Μέσερσιτ που είναι εκτός ποσοστώσεων διότι είναι ε, της έχουν εκλεγεί στην Δανία, από τη Δανία. Για το 2012 τώρα γίνεται, έχει γίνει ένα ε, αίτημα για τις επισκέψεις Ιρλανδία, Κύπρο, ε, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, θα γίνει και μία επίσκεψη στην Καλ, Καλσρούη για το επίσκεψη στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας την, το απόγευμα το απόγευμα ε, αφού ολοκληρωθεί η συνάντηση, η συνεδρίαση της τελευταίας μέρας της Συνόδου στο Στρασβούργο, θα γίνει η συνάντηση. Για τις ακροάσεις του 2012 υπάρχει ένα πρόγραμμα ήδη, βέβαια έχουμε και περιθώρια για περαιτέρω αιτήσει, αλλά επί του παρόντος έχουμε μέθοδ, τις μεθόδους για μία άμεση συμμετοχή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ε, μοντέλο για μια πιο ε, δημοκρατική Ευρώπη. Αυτή είναι η ακρόαση, η μόνη ακρόαση που έχουμε μέχρι στιγμής. Τώρα, εάν υπάρχουν και άλλα αιτήματα, μπορείτε να τα ε, διαβιβάσετε στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Ταρκόφσκι τώρα θα ασχοληθεί με τη διαθεσμική συμφωνία που θα συνοδεύσει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Και θεωρήσαμε ότι δεν είναι ε, σκόπιμο να ορίσουμε έναν εισηγητή για την ε, απαλλαγή για, τον, για την εκτέλεση του προπολογισμού του 2010. Τώρα, σύμφωνα με το άρθρο 50, έχουμε δύο αιτήματα ε, που έχουν υποβληθεί και στη μία έχω απαντήσει γραπτά, στην ε, δεύτερη, τη δεύτερη που μόλις την έλαβα, το δεύτερο μάλλον που μόλις το έλαβα, το έλαβα θα απαντήσω. Θα, απαντή, θα προετοιμάσω μία απάντηση για το ερώτημα το οποίο τέθη που αφορά την ερμηνεία του άρθρου 117. Τώρα, αυτές είναι οι ανακοινώσεις. σχετικά με τα όσα διαμήφθηκαν χτες στην συνάντηση των συντονιστών. Εάν και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, ε, είχαμε αναβάλει για σήμερα την έκθεση που ήταν στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Είναι η κυρία Γκουρμάη. Όχι. Η κυρία Γκουρμάη δεν είναι στην αίθουσα ακόμα, άρα περιμένουμε. Θα συζητήσουμε επομένω τον κώδικα συμπεριφορά των βουλευτών. Όπω ξέρετε, έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ για αυτό το θέμα και πιο συγκεκριμένα και στην προηγούμενη μα συνεδρίαση, αλλά αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και σε αυτή τη ε, συνεδρίαση τη συζήτησή μα. Θα ε, μου επιτρέψετε να συνοψίσω τα όσα έχουμε συζητήσει, τα όσα είπαμε μέχρι τώρα Λοιπόν, όπως ξέρετε, και συνοψίζω τη θέση μου, ε, εν συντομία, μία ομάδα εργασίας έχει συντάξει έναν κώδικα συμπεριφοράς. Αυτή η ομάδα εργασίας έχει διαβιβάσει το αποτέλεσμα της εργασίας των εργασιών της στο Προεδρείο, στην Συνεδρία των Προέδρων και ε, εγκρίθηκε. Βέβαια, ένας κώδικας συμπεριφοράς ήδη υπάρχει σήμερα στο παράρτημα 2 που ισχύει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, σύμφωνα με την πρότασή μου, να, αφορά, να ασχοληθούμε όχι μόνο με το παράρτημα 1, αλλά και κάποια του κανονισμού, αλλά και κάποια άρθρα του κανονισμού του ίδιου το, άρθρο 9, 32, 156 και ενδεχόμενα και το άρθρο 19 ανάλογα με την απόφαση που θα πάρουμε. Αυτό είναι ένα πράγμα. Επίσης, θεωρώ ότι δεν αρχεί να αντικαταστήσουμε το παράρτημα 1, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να τροποποιήσουμε και το άρθρο 9 έτσι ώστε να γίνεται σωστή αναφορά στο παράρτημα. Και αυτό το άρθρο το σημείο 9 είναι τυπικό βέβαια. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Υπάρχουν όμως δύο προβλήματα, ε, τα οποία αφορούν καταρχάς τις παραλήψεις του κώδικα συμπεριφοράς έτσι όπως έχει συνταχθεί από την ομάδα εργασίας, ε, παραλήψεις που ήδη αναφέρονται όμως στον υπάρχοντα κώδικα συμπεριφοράς και ε, είναι ας πούμε η ανάγκη από πλευράς ε, μάλλον να αναφέρονται να αναφέρονται από τους κοσμήτορες ε, τα χρήματα τα οποία ανατίθεται σε διάφορες επιτροπές. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι λογικό να παραμείνει η υποχρέωση αυτή όχι στον κώδικα συμπεριφορά αναγκαστικά, αλλά να συμπεριληφθεί στο άρθρο 32 του κανονισμού, εκεί που αναφερόμαστε στις διακομματικές ομάδες. Το δεύτερο θέμα αφορά τις κυρώσεις. Ο κώδικας συμπεριφοράς προβλέπει πέντε ειδών κυρώσεις, που, ε, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι αυτές που προβλέπει ο κανονισμός στα άρθρα 153 και άρθρα 156. Όμως προσθέτει και μία έκτη κύρωση που είναι η ανάκληση ε, της ε, εντολής ε, που έχει δοθεί σε κάποιον για να συντάξει μια έκθεση. Ανακαλείται ως συντάκτης. Λοιπόν, θεωρούμε ότι οι κυρώσεις θα έπρεπε να αναφέρονται στον κανονισμό των ίδιων. Δηλαδή δεν θα πρέπει οι κυρώσεις να αναφέρονται ε, στο κώδικα συμπεριφοράς, δηλαδή στο παράρτημα 1, αλλά στο άρθρο 153. Αν συμβεί αυτό όμως, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στον κατάλογο των κυρώσεων και αυτή η έκτη ποινή, αν θέλετε, που είναι η ανάκληση του, της του συντάκτη. Κατά την άποψή μου, το άρθρο 19 δεν τροποποιείται το άρθρο 19 του κανονισμού, διότι το άρθρο 19 αναφέρεται στην έκπτωση από κάποιο ερετό αξίωμα. Και ο ισχύων ο κώδικας συμπεριφοράς όσον αφορά την, ανά, την έκπτωση και την ανάκληση των αρμοδιοτήτων και από την θέση ενός ερετού ε, ε, άρχοντα τέλος πάντων αναφέρονται στο άρθρο 19 και δεν εδώ δεν εμπίπτει η ποινή κύρωση που αφορά την ανάκληση από τη θέση του, του συντάκτη. Εδώ η διάσκεψη των Προέδρων ή μια ειδική πλειοψηφία αρκεί για να, πά, για να ληφθεί μια απόφαση που θα ε, επικυρώσει την απόφαση της ε, Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Επομένως, εάν θέλουμε να αναφερθούμε στις ποινές ε, του άρθρου 153 χωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε προστίκη για την ανάκληση της θέσης του, εισηγητή, του συντάκτη, συγγνώμη, του εισηγητή, ε, μπορούμε να ερμηνεύσουμε το άρθρο 19 και να, το, να προσθέσουμε εδώ ότι αρετό αξίωμα ε, σημαίνει και η, η θέση του συντάκτη. Άρα και για το, ε, και για τον να ε, στα, ε, πάψει να είναι κάποιο συντάκτη, εισηγητή συγγνώμη, μια έκθεση, χρειάζεται η ειδική πλειοψηφία ή όλη η διαδικασία τέλο πάντων που απαιτείται και για την έκπτωση από κάποιο ερετό αξίωμα. Αυτές είναι οι απόψει της ομάδα εργασία. Η ομάδα εργασία για αυτή τη νέα κύρωση προβλέπει ο πρόεδρος να αναθέτει στην διάσκεψη των προέδρων, στη διάσκεψη των προέδρων, ναι, στη διάσκεψη των προέδρων, το θέμα. Δεν λέει όμως ποιος αποφασίζει. Αποφασίζει η διάσκεψη των προέδρων. Αυτό όμως η ομάδα εργασίας δεν το λέει. Ή η, η διαβίβαση στην διάσκεψη των προέδρων ε, συνεπάγεται και εφαρμογή του άρθρου 19. Το περίεργο είναι ότι το κείμενο το οποίο έχει διαβιβάσει η ομάδα εργασίας αναφέρει το άρθρο 19 όσον αφορά την αναστολή ή την έκπτωση από ένα αιρετό αξίωμα ε, που είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στο 19, αντιπρόεδρος, ο Κοσμήτορας, ε, πρόεδρος ή αντιπρόεδρος Επιτροπής. Δεν αναφέρει τίποτε όμως για τη νέα κύρωση που είναι η αναστολή από την θέση του εισηγητή μιας έκθεσης. Άρα αυτή η διαφορά τι σημαίνει. Παραμένει σε εν κενό το, το θέμα του ποιος θα πρέπει να επιβάλλει την κύρωση αυτή. Και εγώ προτείνω να πούμε, για να, αναπλουστεύσουμε τα πράγματα, ότι το άρθρο, να προσθέσουμε στο άρθρο 19 μια διάταξη που να λέει ότι ε, για, την, για τον κανονισμό αυτό ο ορισμός ενός ε, εισηγητή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή του άρθρου 19. Θεωρείται δηλαδή σαν ερετό αξίωμα. Εγώ από την άλλη πλευρά θεωρώ όμως ότι επιβαρύνεται η διαδικασία. Δηλαδή για τα ερετά αξιώματα ισχύει το άρθρο 19. Όμως και κάποιες ε, θέσεις και κάποιες θέσεις για τους συζητές λοιπά ορίζονται από τις επιτροπές. Άρα θα πρέπει η διάσκεψη των Προεδρών να, να αναθέσει στις αρμόδιες επιτροπές το, την αρμοδιότητα για να ε, αναστείλει την, ε, τις αρμοδιότητες εισηγητή από κάποιον. Να αφαιρέσει, αν θέλετε, το, τη θέση του εισηγητή από κάποιον. Από κάποιον στον οποίο έχει αναθέσει η ίδια η Επιτροπή, βέβαια, την, τον ρόλο του εισηγητή. Λοιπόν, επομένως υπάρχουν, ε, υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία, εκτός από κάποιες ε, διορθώσεις, αν θέλετε, και ένα θέμα μόνο παραμένει σε εκκρεμότητα, είναι ποιος θα πρέπει να αποφασίσει για την αναστολή ε, από την θέση του εισηγητή. Ακούστηκαν πολλές απόψεις σας, τις οποίες έχω καταγράψει. Δεν πρόκειται όμως να τις αναφέρω, γιατί ε, δεν θα έχουμε το απαραίτητο χρόνο. Ο κύριος Νταφ ζήτησε το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με την προσέγγιση, προσέγγιση σας σε ό,τι αφορά την, ε, τη μεταρρύθμιση του κώδικα και του κανονισμού. Έχω κάνει και στο παρελθόν ε, στις προηγούμενες συζητήσεις σχετικά σχόλια και θα καταθέσω διάφορες ε, τροπολογίες για να πετύχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια στο όλο εγχείρημα το οποίο θεωρώ ότι δεν το πετύχε η ομάδα εργασίας παρά το γεγονός ότι εργάστηκε πολύ σκληρά και μάλιστα επί σειρά μηνών. Δεν νομίζω ότι έκαναν πολύ καλή δουλειά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αλλά Γι' αυτό έχουμε και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Δύο-τρία θέματα τώρα να θίξω. Στην, ε, στο άρθρο 4, τροπολογία 9. Νομίζω ότι την υποπαράγραφο C θα πρέπει να καταστεί σαφές, απόλυτα σαφές, ότι μιλάμε για κανονικές αμοιβόμενες δραστηριότητες για να τονίσουμε την αντίθεση με το ε, το ή, όπου μιλάμε για περιστασιακές ε, αμοιβόμενες ε, δραστηριότητες. Και αν συμφωνείτε με την ερμηνεία μου ως προς αυτό, θα προτείνω μία τροπολογία που θα ορίζει ακριβώς αυτό και λίγο παρακάτω. Στο άρθρο αυτό γίνεται λόγος στην υποπαράγραφο H, ήτα. Νομίζω ότι μιλάμε για επενδύσεις και ε, εισοδήματα από επενδύσεις, δηλαδή μερίσματα από αξιόγραφα, μετοχές και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η δεύτερη παράγραφος όπου γίνεται λόγος για τακτικά εισοδήματα προκαλεί μεγάλη σύγχυση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε σε εισοδήματα, έσοδα από επενδύσεις, τα οποία μπορεί να είναι μεν τακτικά, αλλά μπορεί να είναι και περιστασιακά. Όπως ξέρουμε, οι μετοχές μπορεί να ανέβουν και να κατέβουν σε αξία. Άρα, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει καταρχάς να διευκρινιστεί στο σχέδιο. Ύστερα, στην, ε, στο άρθρο 5, στην αρχή περίπου του άρθρου, στη δεύτερη παράγραφο, σε ό,τι αφορά τα έσοδα από επενδύσεις λοιπόν σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τακτικά έσοδα. Άρα, στο άρθρο 5 τώρα, τροπολογία 10, το συζητήσαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Θα ήθελα όμως να ξέρω αν ο εισηγητής θα καταθέσει οποιαδήποτε τροπολογία. γιατί το να μείνει κανείς ε, σε ένα ξενοδοχείο 4-5 αστέρων όπως το Σοφιτέλ μπορεί να κοστίσει και 200 επιπλέον ευρώ. Τι λέμε δηλαδή, ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου δεν επιτρέπεται να αποδεχτούν την επιστροφή τέτοιων εξόδων διαμονής. Κατά την επίσκεψή τους ε, για τη συμμετοχή σε ένα συνέδριο ή κάτι τέτοιο. Αυτό θεωρώ την ανοησία. Και ειλικρινά αμφιβάλλω και αμφισβητώ το κατά πόσον το άρθρο 5 έχει οποιοδήποτε όφελος. Νομίζω ότι μπορούμε να, να πάρουμε ένα, μια καλύτερη διατύπωση από τον κώδικα διοντολογία της Επιτροπής, αλλά να σκεφτούμε κατά πόσο οι βουλευτές οι οποίοι, δεν, οι βουλευτές οι οποίοι δεν είναι μέλος του εκτελεστικού θα πρέπει να υπόκεινται τις ίδιες περιορισμούς όπως η Επιτροπή. Στο άρθρο 7, τελευταίο σημείο, τροπολογία 12, Νομίζω ότι στο τέλος θα πρέπει να προσταθεί μια νέα υποπαράγραφος 6 για να ορίσουμε ότι η συμβουλευτική αυτή επιτροπή θα δημοσιεύει μια αιτήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο για να τηρούμε ένα μητρό αυτό μάλλον θα δημιουργήσει προηγούμενα. Αν το κάνουμε αυτό, δεν πρόκειται να διευκρινίσουμε με καλύτερο τρόπο τα καθήκοντα της ε, Επιτροπής. Νομίζω ότι δεν θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τις πρακτικές μας εμπειρίες και να δημοσιεύονται όλα αυτά προκειμένου το Κοινοβούλιο να εξεγάγει τα απαραίτητα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα... Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα καλά, κύριε Ντάφ, μια διευκρίνηση. Όταν αναφέρεστε στην τροπολογία 9, στην τροπολογία 9 λέτε ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε, αν κατάλαβα καλά, και την αναφορά σε περιστασιακές δραστηριότητες. Δεν είμαι βέβαιος αν κατάλαβα, γιατί ούτως ή άλλως στην ε, τροπολογία 9 στο ε οποιαδήποτε περιστασιακή αμοιβόμενη εξωτερική δραστηριότητα περιλαμβανομένων συγγραφικής δραστηριότητας, δεκτικού έργου κλπ. Επομένως η περιστασιακότητα εδώ αναφέρεται ή κάνω λάθος, μήπως αναφερόσασταν σε κάτι άλλο. No, there are, I think, three... Νομίζω ότι υπάρχουν τρία είδη εσόδων τα οποία μπορεί να έχει ένας βουλευτής. Πέρα από τον κοινοβουλευτικό του μισθό. Καταρχάς αναφέρεται στο γάμα, στο σι, στην υποπαράγραφο γάμα. Αυτό ασφαλώς σημαίνει οποιαδήποτε, οποιασδήποτε αμοιβόμενε αμοιβόμενες ε, δραστηριότητες. Στο ε, στο ε, γίνεται αναφορά σε περιστασιακές τέτοιες δραστηριότητες, μη τακτικές δραστηριότητες αμοιβόμενες. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει σαφέστατη αυτή η αντίθεση. Στην τρίτη περίπτωση τώρα, στην υποπαράγραφο γίνεται λόγος για επενδύσεις και για έσοδα από επενδύσεις. Μερίσματα, έσοδα από αποτομίευση. Αυτό θα ήθελα να το ορίσουμε καλύτερα, γιατί αν σωστά ερμηνεύω το νόημα όλων αυτών, θα πρέπει να γίνει καλύτερη διάκριση από ό,τι γίνεται στο παρόν σχέδιο. Αν κάνω λάθος δε, τι να σας πω, δεν καταλαβαίνω σε καμία περίπτωση τι νόημα έχει το άρθρο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρτιν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Τρεις παρατηρήσεις μόνο. Καταρχάς, αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Νταφ ε, προς το τέλος της παρέμβασής του για τις συμβουλευτικές επιτροπές. Έχω κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσον ε, η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να δώσει συμβουλές αλλά και ερμηνείες στα μέλη και ε, σε κατοπινό στάδιο να είναι και δικαστής και να δει αν εφαρμόζεται σωστά ο κώδικας διοντολογίας. Είναι σαν να με δύο διαφορετικούς κανόνες, αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι έτσι είναι και θα πρέπει να το δεχτούμε. Στην τροπολογία 12 νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε στο σημείο 3 ότι θα πρέπει να δίνονται συμβουλές ε, ε, με εμπιστευτικό χαρακτήρα. Αυτό δεν είναι αντίθετο σε αυτό που προτείνει ο κύριος Νταφ για την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία μπορεί να δημοσιεύεται για τις γενικότερες συμβουλές που έχουν δοθεί, αλλά δεν χρειάζεται να δίνονται λεπτομέρειες για το ποιο ρώτησε τι και γιατί το ρώτησε. Τώρα, για τις μικτές ομάδες ε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Η ε, πρόθεση της διάσκεψης των Προέδρων είναι σαφής, θέλει να ενισχύσει τον κώδικα διοντολογίας και νομίζω ότι ορθώς το διορθώνεται. Για τις κυρώσεις τώρα. αυτή για τους εισηγητές είναι δύσκολη και για μένα. Καταλαβαίνω ποιο είναι το σκεπτικό σας και προτείνετε να χρησιμοποιείτε το άρθρο 19. Θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 19 με την παραλλαγή στην οποία αναφέρεστε. Αντί να απαιτείτε πλειοψηφία 3 πέμπτα στην Ολομέλεια, θα μπορούσαμε να έχουμε μια ξεχωριστή φράση που να λέει ότι για τους εισηγητές ισχύει η ίδια η διαδικασία μόνο που απαιτούνται τρία πέμπτα της αρμόδιας επιτροπής για να αφαιρεθεί ο ρόλος του εισηγητή από κάποιον. Ε, ώστε να μην υπάρχει και πρόβλημα με τις επιτροπές, διότι κατά πάσα πιθανότητα και η επιτροπή θα μπορεί να κρίνει καλύτερα εάν υπήρξε επιρροή από εμπορικά ή άλλες μορφές οικονομικά συμφέροντα για τον εισηγητή. Κατά τα άλλα, εγώ συμφωνώ απολύτως με την προσέγγιση που έχετε κύριε Πρόεδρε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και εγώ, όπως και ο Άντριου, με ανησυχεί το άρθρο 5. Τίθεται θέμα του πόσο συγκεκριμένοι θέλει να είμαστε και πόση ευελιξία χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις. Γι' αυτό και συμφωνώ να υπάρχει μία έκθεση που θα δημιουργεί και κάποιο προηγούμενο, γιατί υπάρχει διαφορά από το να προσκληθεί κάποιο σε ένα ε, συνέδριο και να διανυκτερεύσει σε ένα ξενοδοχείο, από το να προσκληθεί σε διακοπέ πολυτελεία. Γιατί αυτό φυσικά δεν μπορούμε να το βάλουμε στον κώδικα διοντολογία. Και άλλο να δεχτεί κάποιο ένα βιβλίο ως δώρο από μια διάσκεψη που στοιχίζει 150 ευρώ. On, uh, on article 5, we keep... Στο άρθρο 5 τώρα, αν διατηρήσουμε τα θέματα όσα έχουν, θα πρέπει να σκεφτούμε εάν θα πρέπει να αντιγράψουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπε και ο Άντρου, αλλά καλό θα ήταν να ναι, έχουμε και αυτή την έκθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις για να ε, ξέρουμε τι γίνεται και να λέμε ότι σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να γίνει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό και σε γενικές γραμμές συμφωνώ και με την προσέγγιση του Προέδρου, την οποία και ε, δέχομαι. Ο κύριος Καζίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, να επαναλάβω και εγώ όσα είπαν οι άλλοι, τα οποία με βρίσκουν σύμφωνοι, σύμφωνο. Ιδιαίτερα αυτά που είπε ο κύριος Ντάφ και ο κύριος Μάρτιν. Θεωρώ πάντως ότι θα πρέπει στο άρθρο 3 να υπάρχει κάποια χρονική περίοδος, γιατί είχα προτείνει η Εξεταστική Επιτροπή, η Συμβουλευτική Επιτροπή να απαντάει εντό 30 ημερών. Να μην υπάρχει δηλαδή απεριόριστο ε, περιθώριο σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση τη Επιτροπή αυτή. Να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη υποχρέωση. Εγώ θα ήμουν υπέρ όχι μια ετήσια έκθεση, αλλά ενό διαρκού μητρώου, γιατί νομίζω ότι θα, θα δημιουργηθεί ένα σώμα προέδρων. Θεωρώ ότι σωστό λοιπόν είναι να καταγράφονται όλα αυτά και η διαβούλευση από τους βουλευτές να μπορεί να γίνεται ανα πάσα στιγμή η εξέταση των, του Μητρώου αυτού. Νομίζω ότι θα πρέπει η Επιτροπή αυτή, αν θέλουμε να είναι νόμιμη και να έχει νομιμοποίηση, όχι να διορίζεται, αλλά να εκλέγεται. Ε, Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Σημειώνω λοιπόν ότι υπάρχει σε γενικές γραμμές συνένεση για την έκθεσή μου οι παρατηρήσεις που κάνατε θα μπορούσαν να διατυπωθούν μέσω τροπολογιών, τις οποίες σας παρακαλώ και να καταθέσετε. Ακόμα και σε περιπτώσεις που θεωρώ ότι κάποιες τροπολογίες σας ε, θα πρέπει να γίνουν δεκτά, δεν θα ε, τις καταθέσω εγώ ως τροπολογία. Εγώ θα κάνω μία τροπολογία μόνο για την ε, ανάκληση του εισηγητή, ε, αλλά ε, για τις υπόλοιπες παρατηρήσεις σας, κατ' θα πρέπει να καταθέσετε τροπολογία και γραπτός θα μπορέσουμε να τις ε, αξιολογήσουμε καλύτερα. Κάποιες από αυτές με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά δεν θα τις ε, καταθέσω εγώ ως τροπολογία. 27 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Νομίζω ούτως ή άλλως ότι έχει οριμάσει πλέον η συζήτηση, δεν υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε την προθεσμία αυτή και επομένως ε, τη συζήτηση για το θέμα αυτό και μπορούμε ε, possiamo Θα έλεγα λοιπόν πριν ε, ψηφίσουμε να περάσουμε στην έκθεση του κυρίου Τρασκόσκη για την Κροατία. Έχετε το λόγο, μπορείτε να μας πείτε τα της Κροατίας. Βασικά, πρέπει να ετοιμάσουμε μια γνωμοδότηση για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα. Και εμείς καθήκον έχουμε να ε, μιλήσουμε για τη συνταγματική κύρωση της ε, διαδικασίας αυτής. Δεν ε, μιλάμε στη γνωμοδότηση αυτή για την φιλοσοφία της διεύρυνσης, ασχολούμαστε αποκλειστικώς και μόνο με την Κροατία. Βέβαια υπάρχουν ένα-δύο παράγραφοι στην αρχή που αναφέρονται στην ε, διαδικασία ένταξης αυτή καθ' αυτή. Ε, αποφάσισα να ξεκινήσω από τα θετικά στοιχεία. Πάντα είναι υποσυζήτηση το θέμα της διεύρυνσης και οι επιπτώσεις της, αλλά είμαι πεπισμένος ότι η διεύρυνση ε, πηγαίνει από κοινού με την ε, συνταγματική και θεσμική μεταρρύθμιση και μάλιστα δρά και καταλητικά για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο συνταγματικό σύστημα. Δεν ε, επιδρά αρνητικά λοιπόν στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει, ίσα ίσα μας βοηθά να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Επιπλέον θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά από την ε, έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας, υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, υπάρχει και ρήτρα διαφύλαξης για τη σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι λοιπόν στην αρχή στη διαδικασία της κύρωσης, υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν συνεχώς ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις της διεύρυνσης, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, Αναφερόμαστε επίσης στο θέμα του δημοψηφίσματος στην Κροατία και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας είναι το θέμα της νέας σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο μπορεί να επιληθεί βάσει της συνθήκης. Ε, τέλος, καλούνται τα κράτη-μέλη να περάσουν ε, στη διαδικασία κύρωσης της ε, ε, ε, με την Κροατία χωρίς να το περιπλάξουν με άλλε διαδικασίες για να μην υπάρχει περαιτέρω καθυστέρηση στην ημερομηνία ένταξης. Ε, βρισκόμαστε άλλωστε σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις ουσιαστικέ εργασίες τη Ευρωπαϊκής Ένωση. ανεξάρτητα από τα προβλήματα και είμαστε ανοιχτή σε νέε διευρύνσει, ιδίω σε χώρε οι οποίε είναι έτοιμε και έχουν ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει και αυτό ισχύει φυσικά για την Κροατία. Αποτελεί θετική ένδειξη και νομίζω ότι αυτό το θετικό μήνυμα θα πρέπει να αποσταλεί και από την Επιτροπή μας αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Αυτά λοιπόν είναι η εισαγωγή. Ο κύριος Ντάφ. Could I Θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή πότε θεωρεί ότι θα υπογραφεί η συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας. Και κατά δεύτερον στην παράγραφο 7 αναφέρεται ότι η επικύρωση δεν θα πρέπει να συνδεθεί με τις διαδικασίες επικύρωσης του Ιρλανδικού πρωτοκόλου, του Τσεχικού πρωτοκόλου. Νομίζω όμως ότι υπάρχει πολιτική απόφαση, απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι επρόκειτο να υπάρξει τέτοια σύνδεση, δηλαδή να υπάρχει μια παράλληλη αλλά ενιαία διαδικασία επικύρωσης τους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει αυτό να αποτυπώνεται στην ε, διατύπωση της ε, γνωματότησης. Η απόφαση δηλαδή αυτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υποδεικνύοντας παράλληλα ότι ενδεχομένως να υπάρξει αντίκτυπος και μάλιστα μη επιθυμητός από το τσεχικό και το ιρλανδικό πρωτόκολλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε φάση που καταρτίζουμε διάφορες εκθέσεις από αυτού. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ να ρωτήσω κάτι προς διευκρίνηση για την παράγραφο 7 και εγώ αυτές οι συζητήσεις για τις άλλες διαδικασίες επικύρωσης από ποιον γίνονται και σε ποιο πλαίσιο από εθνικά κοινοβούλια θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη σαφήνεια. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Εγώ μπορεί να αφαιρέθηκα, ζητώ συγγνώμη. Ε, θα ήθελα να κατανοήσω ποια είναι η άποψη του εισηγητή για τις έδρες στο Κοινοβούλιο μετά την ένταξη της Κροατίας. Ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο σαφής η παραγραφός 7, διότι αναφέρεται σε δύο διαφορετικά πράγματα και καλώς ε, μου το επισημαίνετε διότι υπάρχει άποψη ε, κάποιων κρατών μελών ότι η ένταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από διαδικασία κύρωσης στα κράτη-μέλη και αυτό είναι ανάθεμα για μας στην Επιτροπή και φυσικά υπάρχει και το θέμα των επιπλέον πρωτοκόλων και να μην ε, έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση. Θα πρέπει ίσως να το διευκρινίσω για να μην δημιουργεί σύγχυση. Ο κύριος Σέπφλιν έχει δίκιο. Ε, είτε το ένα είτε το άλλο θα εξετάσουμε. Θα προσπαθήσω να είναι λίγο σαφέστερη διατύπωση. Όσον αφορά τώρα την ε, υπογραφή της ε, συνθήκης προσχώρησης, η Πολωνική Προεδρία ενδιαφέρεται να υπογραφεί τώρα, στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, πριν ολοκληρωθεί η Πολωνική Προεδρία και φαίνεται ότι θα το καταφέρουμε. Όσον αφορά τώρα τη σύνθεση του Κοινοβουλίου, Η παράγραφος 6 νομίζω απαντά. Αν χρειάζεται οποιαδήποτε διευκρίνηση ε, θα εξετάσω αν μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο σαφείς. Όσο έχει όμως αυτή τη στιγμή ε, είναι αυτό που ισχύει στη συνθήκη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλό το κείμενο. Θα προσπαθήσω να διατυπώσω λίγο την παράγραφο αυτό. 7 ε, με, τα χαρά. Υπάρχουν άλλε παρεμβάσει. Πριν Α, ζητώ συγγνώμη. Κάνατε κάποιες παρατηρήσεις, όχι πολλές, αλλά κάνατε. Πρέπει να, ρωτήσουμε, να ορίσουμε την, την θεσμία την υποβολή τροπολογιών. Η Επιτροπή ΑΦΕΤ θα γνωμοδοτήσει για την έκθεση Σβόποντα στις 14 Νοεμβρίου, άρα εμείς θα πρέπει να το συζητήσουμε στις 24 Οκτωβρίου. Άρα 5η 13 Οκτωβρίου, μεσημέρι, ορίζεται 13 οκτωβριου μέση ημέρη, οριζεται η προθεσμια για την υποβολή των τροπολογιών, εάν ο εισηγητή σε συμφωνήσει. Δηλαδή, 24 Οκτωβρίου η ψηφοφορία, 13 Οκτωβρίου στι 12 η ώρα η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Προτείνω επομένω τώρα να προχωρήσουμε την, ε, σύμφωνα με την ε, ημερήσια διάταξη για, την, ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, έκθεση Τσαρκσκόφσκι. Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών, το σημείο 13 της ημερησίας διάταξης. Όπως θυμάμαι από τα μαθήματα που έκανα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ε, ένας από τους καλύτερους ορισμούς ήταν ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ένας κινούμενος στόχος. Και το συνειδητοποίησαμε αυτό με την οικονομική διακυβέρνηση και το ε, ευρωπαϊκό εξάμεινο. Είχαμε μία έκθεση της κυρίας Περβόνς, Περές, ε, υποβάλαμε, υποβλήθηκαν τροπολογίες, καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο ορίζει πολύ πιο συγκεκριμένα το θεσμικό ρόλο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μέσω των γνωμοδοτήσεών μας, πολλές φορές και τροπολογιών επίσης ε, και γνωμοδοτήσεων που καταλήγουν σε συμβαστικές τροπολογίες, περνούν, αλλά θα πρέπει κάπως να είμαστε πιο συγκεκριμένοι διότι στην έκθεση της κυρίας Περές ο θεσμικός ρόλος του, του Κοινοβουλίου ορίζεται σαφέστερα. Στην ε, Επιτροπή Έκον, στην έκθεση της Επιτροπής Έκονο ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που ασχολείται με την, ε, που προβλέπει τη δημιουργία μιας υποεπιτροπής μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής ΕΚΟΝ και που θα αποτελείται από μέλη που προέρχονται από την Ευρωζώνη. Αυτά είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Αυτό το θέμα είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, αλλά για μας αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις συνθήκες, άρα θα πρέπει να διαγραφεί αυτή η ιδέα όσο πιο γρήγορα. Επομένως, τι θα κάνω. Θα υποβάλω αυτές τις ε, συμβαστικές τροπολογίες στους συντονιστές και θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε αυτό τον ε, κινούμενο στόχο, κυρίως για τα θέματα που μας αφορούν, δηλαδή για το θεσμικό πλαίσιο. Και αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες θα προσπαθήσουμε να γίνουν πιο συγκεκριμένες και να είμαστε και πιο κοντά στα όσα προτείνει η κυρία Περές για τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε η γνωμοδότησή μας να είναι ενημερωμένη και να λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές που προτείνει η κυρία Περές. Και η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών έχει παραταθεί νομίζω. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τις ημερομηνίε. Γιατί θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η γνωμοδότηση έχει ενημερωθεί και ευθυγραμμίζεται με αυτά τα οποία προτείνει η κυρία Περές. Η προθεσμία για την ε, υποβολή των ε, τροπολογιών έχει περάσει 5 Οκτωβρίου και νομίζω ότι υποβλήθηκε μονάχα και μία τροπολογία από, από εσά. Δεν ξέρω εάν μπορούν να υποβληθούν περαιτέρω συμβαστικέ τροπολογίε τώρα, αλλά η προθεσμία έχει περάσει και ορίστηκε η ημεροπροθεσμία. Τελείωσε. Πρέπει να περάσουμε στην ψηφοφορία στις 24 Οκτωβρίου για να είμαστε σε θέση να παρέμβουμε ε, την κατάλληλη στιγμή. Ε, Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Και μετά ο κύριος Νταφ. Ναι κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα είναι ότι εμείς είχαμε ξανανοίξει την ε, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, εκτός και αν κάνω λάθος, αλλά δεν ε, κατατέθησαν νέες τροπολογίες, γιατί δεν έφτασε εγκαίρως στο νέο κείμενο για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Είχε ξανανοίξει προθεσμία για να αντιδράσουμε στο νέο κείμενο. Δύο πράγματα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε. Ή να ξανανοίξουμε την προθεσμία για την ε, τροπολογία, ε, κατάθεση τροπολογιών, συγγνώμη, ή μαζί με τους ε, σκιώδεις να ετοιμάσουμε κάποιες τροπολογίες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να εξετάσουμε και τη διεύρυνση του, του θέματος της έκθεσης της κυρίας Μπερές. Ένα πράγμα να πω, η υποεπιτροπή είναι βεβαίως κάτι διαφορετικό γιατί υπάρχει διάκριση για τα μέλη του Κοινοβουλίου όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου. Θεωρώ όμως ότι το άρθρο 26 θα έπρεπε να διευκρινίζει ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίσει την Ολομέλεια για όλους τους κανονισμούς που υιοθετούνται βάσει της διαδικασίας του 136 ή ό,τι ε, υιοθετείται βάσει του 121.6, δηλαδή οικονομικοί κανονισμοί που ε, ε, υιοθετούνται από το Συμβούλιο στο 17 και το Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από τη συνθήκη και δεν αποτελεί πρόβλημα και δεν δημιουργεί κάποια συμμετρία στην ε, ε, σύνθεση του Συμβουλίου ή του Κοινοβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση θα είμαστε κατά τη δημιουργία μια υποεπιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν μόνο τα μέλη τη Ευρωζώνη. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το εξετάσουμε λίγο περαιτέρω. Θα δω και τι πρόταση θα κάνει ο συνάδελφος ε, Τρασκόφσκι αν θεωρεί ότι πρέπει να παρατείνουμε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ή να παρουσιάσουμε ε, νέες τροπολογίες σε συνεργασία με τους κοιόδης. Ο κύριος Νταφ. Ναι. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα ο εισηγητής με τους κοιόδης εισηγητές να προσπαθήσουν να ετοιμάσουν μια συμβαστική πρόταση. Η έκθεση της κυρίας Μπερές άλλαξε κατεύθυνση από τότε που ξεκίνησε πριν από πολύ καιρό και και βεβαίως ε, είναι πολύ σημαντικό το συνταγματικό ερώτημα το οποίο θέτει. Θα δημιουργηθεί και προηγούμενο. Εάν παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, η πείρα καταδεικνύει ότι αν εμείς ως Κοινοβούλιο αρχίσουμε να συμφωνούμε στον κατακαιρματισμό της συνοχής του Κοινοβουλίου θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθουμε στην πρώτη κατάσταση. Δεύτερον, η κυρία Μπερές προσπαθεί να δώσει εντολές ουσιαστικά στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου όταν πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω απόφασης Επιτροπής δηλαδή ότι η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, θα έχει την εξουσία να δίνει εντολή στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Και νομίζω ότι πρέπει να τεθεί ένας φραγμός εδώ. Μόνον η Ολομέλεια μπορεί να δώσει εντολή στον Πρόεδρο. Κύριε Τρασκόφσκι, μήπως θέλετε να απαντήσετε. Πρέπει να μας πείτε, συν τις άλλες, αν θεωρείτε ότι πρέπει να παραταθεί η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι πολύ σύντομη η προθεσμία. 13 Οκτωβρίου, αύριο μεθαύριο δηλαδή. Ή αν αντί να παρατείνουμε την προθεσμία να κάνουμε συμβαστικές προτάσεις. Why was it confusing a Μου προκαλέστηκε κάποια σύγχυση γιατί για κάποιες ε, οι ιδέες σε ό,τι αφορά τις ε, συνεδριάσεις, όλα αυτά ε, τα αναφέρουμε στην έκθεση. Δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί πολύ απλά ε, τροποποιούμε τις ήδη υπάρχουσες συμβαστικές τροπολογίες αλλά σε ό,τι αφορά τα νέα θέματα, για παράδειγμα την νέα υποεπιτροπή και υπάρχει και ένα νέο θέμα, νομίζω ότι η Επιτροπή Νομισματικών Οικονομικών Υποθέσεων ε, υπερβάλλει κάπως όταν αναφέρει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το καθεξής. Νομίζω ότι πρόκειται για μια σύγχυση ε, των συζητήσεων. Αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να γίνει στη δική μας Επιτροπή. Ξέρουμε πόσο ευαίσθητα άλλα είναι τα θέματα αυτά. Άρα, ουσιαστικά, θα πρέπει να προετοιμάσουμε νέα, νέους συμβιβασμούς, νέες συμβαστικές τροπολογίες, οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Άρα, θα προσπαθήσω να προετοιμάσω αυτές τις νέες συμβαστικές τροπολογίες για να έχουμε κάτι να δουλέψουμε και μετά θα δουλέψουμε με τους σκιώδεις εισηγητές από αυτών των ε, τροπολογιών. Και αν θέλουν οι σκιώδεις να προσθέσουν κάτι, προφανώς και θα το δεχτώ. Γιατί είναι κάπως ε, περίεργες ε, οι συνθήκες στις οποίες θα πρέπει να κατακτήσουμε την έκθεση. Προφανώς έχουν αλλάξει και έχει αλλάξει και η κατάσταση. Και προφανώς και η γνωμοτότηση θα πρέπει να αποτυπώνει όλα αυτά τα καινούργια στοιχεία τα οποία προέβαλε και η Περβάνος Περέσα. Μία πάρα πολύ μικρή διευκρίνηση. Δεν έχω αντίρρηση για την διαδικασία πρώτη ο εισηγητής. Βέβαια, εάν υπάρξουν προτάσεις ε, τελείως διαφορετικές από αυτές που, έχουν, που έχουμε μέχρι στιγμής. Θα ε, ζητήσουμε και την συνεργασία της Επιτροπής, αλλά νομίζω ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά. Τώρα σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Ντάφα για τα θέματα τα οποία θίγει η έκθεση Περέση, για τα θεσμικά θέματα, πιστεύω ότι θα έπρεπε να τονίσουμε περισσότερο την ανάγκη η Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων να ασχοληθεί άμεσα με τα τόσα σοβαρά θέματα όπως είναι η οικονομική ε, διακυβέρνηση του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλώς και μόνο να αντιδρά στις προτάσεις των άλλων θεσμικών οργάνων και να μην λειτουργούμε σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που μας έχει δώσει η συνθήκη εφόσον εκπροσωπούμε ε, τους ψηφοφόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είμαστε αιρετοί άρχοντες, αν θέλετε, αιρετοί... Ε, μας έχουν εκλέξει οι, οι Ευρωπαίοι πολίτες για να κάνουμε το καθήκον μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν λέω ότι θα πρέπει να το κάνουμε τώρα, αλλά θα πρέπει να μπει στα σκαριά ε, και μία έκθεση για τις θεσμικές πτυχές της ε, οικονομικής, της οικονομικής διακυβέρνησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάω απλώς και μόνο για τα θεσμικά θέματα, για τις θεσμικές πτυχές του θέματος αυτού. Δηλαδή, είναι περίεργο ο μόνος οργανισμός ο οποίος δεν συμμετέχει στην όλη αυτή τη διαδικασία να είναι η Επιτροπή Θεσμικών ε, Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, λέει ο Πρόεδρος. Το συζητήσαμε χθε στην ε, Επιτροπή των Συντονιστών, στους των συντονιστών και επικράτησε η άποψη ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Επομένως, αποφασίσαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή Μπαρόζο μάλλον να έρθουμε σε επαφή με την Επιτροπή Μπαρόζο και ήδη έχουμε ξεκινήσει τις επαφές. Τώρα, εάν Θέλει ο κύριος Γκουαλτιέρη να παρέμβει ξανά, εντάξει, ίσως τώρα, ή να παρέμβουμε και εμείς εν γέννη, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν, κανείς άλλος δεν ζητάει το λόγο, ο κύριος Τσαρκόφσκι. Πρόεδρε, θα πρέπει να κοιτάξουμε τα πιο ευρεία θέματα, τα οποία συζήτησαμε και χτες. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε με τον Παρόζο και προφανώς θα πρέπει να υπάρξει και μια έκθεση γιατί δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα στην νομοδοτηση ωστοσο Ωστόσο θεωρώ ότι ένα-δύο θέματα τα πιο σημαντικά θα πρέπει να τα διαπραγματευτούμε στις ε, συμβαστικές τροπολογίες, να δώσουμε μια κατεύθυνση τουλάχιστον, αλλά με πιο ευρύ τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά σε μια έκθεση. Να ακούσουμε όμως πρώτα τον Παρόσο, μήπως μας διαφωτίσει και όπως είπε και ο πρόεδρος του συντονιστές χθες, να δούμε πώς θα συνεχίσει η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νταφ. Οι συντονιστές ε, το συζήτησαν αυτό χτες. Αναγνωρίζουμε ασφαλώς ότι βρισκόμαστε σε μια ομοσπονδιακή στιγμή, όπως θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε. Και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο εσωτερικό, στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο δημιουργίας οικονομικής διακυβέρνησης. Υποπτεύομαι ότι μέχρι την επόμενη άνοιξη θα υπάρξει μια σύμβαση και το Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει όλους τους πολιτικούς και πνευματικούς του πόρους για να καταστεί επιτυχές το εγχείρημα αυτό. Ελπίζω ο Πρόεδρος Μπαρόσο να αποτεχτεί την πρόσκληση στην Επιτροπή για ανταλλαγή απόψεων. Μετά τη συνάντηση της 23ης ε, του μηνός. Κι υπάρξει συμφωνία μεταξύ κυρίου Μπαρόσο και κυρίου Φαντρομπάη στη φάση αυτή σε ό,τι αφορά τη σωστή κατεύθυνση και συμφωνία επί της διαδικασίας με την οποία θα πετύχουμε το στόχο μας αυτό, θα πρέπει να ζητήσουμε από τον πρόεδρο Φαρόμπαϊ να έρθει και αυτός ενώπιόν μας ασφαλώς σε ξεχωριστή περίσταση. Έφνερ. έχει το λόγο. για το σημείο αυτό συμφωνήσαμε χτες για να απευθύνουμε αυτή την πρόσκληση η οποία ελπίζουμε να γίνει σύντομα δεκτή και στη συνέχεια να προβούμε στα επόμενα βήματα. Εγώ προσωπικά το είπα και χτες άλλωστε. Θεωρώ ότι είναι σωστή η πρόταση του συναδέλφου Γκουαλτιέρη να μην περιμένουμε μόνο και να αντιδρούμε μόνο, αλλά σε μια τέτοια κατάσταση η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο γενικά να δημιουργήσει μια δική του εικόνα, να τοποθετηθεί και το ίδιο για να διδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω την πρόταση που έγινε και θα δούμε τι θα αποφασιστεί και στη συζήτηση. Εγώ προσωπικά είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω εκ νέου το θέμα αυτό. Ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορεί κάποια μέλη της Επιτροπής να μην ε, είναι επαρκώς ενημερωμένα για την υπόθεση την οποία συζητάμε. Το Σεπτέμβριο, ο συντονιστής των σοσιαλιστών και δημοκρατών παρουσίασα μία πρόταση προκειμένου η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να εγκρίνει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τις συνταγματικές επιπτώσεις ε, της διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Το συζητήσαμε ένα-δυο φορές στη συνεδριά των συντονιστών. Μέχρι τώρα η πρόταση δεν έχει γίνει πλήρως αποδεκτή. Εγώ λοιπόν ερμηνεύω, δεδομένου ότι είναι παρόντες και αρκετοί από τους συντονιστές που συμμετείχαν χθε στην συνεδρία των συντονιστών, ότι στη χθεσινή συνεδρίαση το γενικότερο πνεύμα και κλίμα ήταν να γίνει αυτή η έκθεση αλλά ότι δεν είχε φτάσει ακόμα η κατάλληλη στιγμή για να ε, εκπονήσουμε την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι από τη σημερινή συζήτηση και από τη δυναμική των απαντήσεων και αυτού του κινούμενου στόχου στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Στρασκόφσκι, ο οποίος ε, ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε συνεχώς προσεκτικοί γιατί υπάρχουν νέες προτάσεις και νέες θέσεις. Ε, προκύπτει σαφώς ότι πρέπει ήδη εμείς εδώ ως Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να εξετάσουμε το θέμα αυτό και να κάνουμε την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Εχθές αποφασίστηκε αυτό που αποφασίστηκε, αλλά εγώ προτείνω, προτρέχοντας λίγο, στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών, να δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα και όχι μόνο το περιεχόμενο. Εχθές σταθήκαμε στο περιεχόμενο, την ανάγκη δηλαδή να σκεφτούμε τα θέματα αυτά. Δεν ε, θεωρήσαμε ότι ήταν επίγον το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με το χρονοδιάγραμμα και να εγκρίνουμε την εκπόνηση αυτή τη έκθεση της πρωτοβουλία. Ναι, το σημειώνω αυτό το είπατε και χθε, ε, σημειώνεται και στα πρακτικά, και εγώ προσωπικώς ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ζήτημα. Το πρόβλημα έγκυται κατ' εμέ στο γεγονός ότι για να παρουσιάσουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας η οποία ε, θα είναι σημαντική διότι δεν μπορεί να είναι απόν το κοινοβούλιο σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Πρέπει να υπάρχουν ιδέε και για να υπάρξουν ιδέε πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα. Ε, αν ακούσουμε λοιπόν τον Παρόζο, θα είναι ίσως χρήσιμο γιατί θα προταθούν σε μας ιδέες προς συζήτηση. Δεν ξέρω ε, αν ε, με προσέχει ο κύριος Γκουαλτιέρη. Μήπως θα έπρεπε πριν αποφασίσουμε να κάνουμε αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας να κάνουμε μια πιο ελεύθερη συζήτηση εμείς εδώ για το θέμα αυτό των ε, θεσμικών ψυχο, πτυχών της ε, οικονομικής διακυβέρνησης χωρίς να ζητήσουμε απευθεία μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για να κατανοήσουμε καλύτερα εμείς τι προβλήματα υπάρχουν και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Ο κύριος Γκολτιέρη. Ναι, θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε στην Επιτροπή αυτή ελεύθερα για αυτό το θέμα, όπως έχουμε ζητήσει και για άλλα θέματα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να δείξει ότι το κοινοβούλιο μας είναι ε, σε θέση να εκφράσει τις δικές του απόψεις και όχι αυτές που εκφράζει ο Μπαρόζο ή ο Βαν Ρομπέι. Όμως, ποιος είναι ο κίνδυνος τον οποίο βλέπω εγώ. Είναι ότι εμείς ε, θα εργαστούμε και το μόνο που θα κάνουμε είναι Απλώς να συμπληρώσουμε την έκθεση έκονο που θα αφορά τα θεσμικά θέματα της ε, οικονομικής διακυβέρνησης. Σε σέβομαι απόλυτα την Επιτροπή έκονο. Όμως τα θεσμικά θέματα είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής των Θεσμικών Θεμάτων. Αυτό το κίνδυνο υπογραμμίζω με την καθυστέρηση αυτή, η έκθεση η οποία θα εγκριθεί στο, στην, στην Ολομέλεια πριν από την ε, ε, διάσκεψη, από τη Σύνοδο Κορυφής ε, του Δεκεμβρίου. Θα είναι η Επιτροπή ΕΚΟΝ και το μόνο που θα κάνουμε εμείς είναι να νομοδοτήσουμε απλώς και μόνο πάνω σε ένα κείμενο το οποίο είναι ήδη παλιό. Άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε ένα ε, χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν θα θέτει στο, στο περιθώριο την Επιτροπή μας, διότι αυτό γίνεται τώρα. Νομίζω ότι η αποδυνάμωση του ευρώ και των θεσμικών υποθέσεων καταδεικνύουν καθημερινά την ανάγκη να μην περιμένουμε. Ο κύριος Μπαρόζο μας έκανε πάρα πολλές προτάσεις για το πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση το καλοκαίρι και νομίζω ότι εμείς ως θεσμός, ως θεσμικό όργανο, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε ο συνάδελφος Καλχέρη. γιατί νομίζω ότι είναι καθήκον μας να εκφραστούμε για το πώς φανταζόμαστε ότι θα προχωρήσουμε και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τον κύριο Μπαρόσο και τον κύριο Φαρόμπαϊ. Πάντα συζητάμε ασφαλώς μαζί τους, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η δουλειά μας και η Επιτροπή μας θα πρέπει να δραματίσει τη σημαντική της, το σημαντικό της ρόλο, να υπογραμμίσουμε ποιες είναι οι δικές μας θέσεις και να μην ε, πάντα γνωμοδοτούμε αποδυναμωμένα σε τοποθετήσεις της Επιτροπής Νομισματικών Υποθέσεων, Οικονομικών Υποθέσεων. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε το έργο μας και να ακολουθήσουμε τις προτάσεις του συναδέλφου κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Πρόεδρε. Χτες δεν ε, ήμουν στη συνεδρίαση των συντονιστών, αλλά νομίζω ότι αυτά που συζητάμε αποτελούν τις βάσεις και τις αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 27 κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν μια κατάσταση όπου οι πολίτες τους αμφιβάλλουν ιδιαίτερα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εμείς ως Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων υποχρεούμαστε να αναλάβουμε πρωτοβουλία και όλες αυτές τις πτυχές να τις ε, συνεισφέρουμε επικοδομητικά στην όλη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτά που είπε ο συνάδελφος Γκατιέρη και οι υπόλοιποι συνάδελφοι υπέρ μιας κοινωνικής πρωτοβουλίας της ε, Επιτροπής μας με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο και νομίζω ότι αποτελεί ένα σημαντικό, μια σημαντική πτυχή που ξεκαθαρίζει ότι ίσως και ως ε, Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων θα πρέπει επί της αρχής να σκεφτούμε τις νέες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα με μια προοπτική για το μέλλον, δηλαδή να κοιτάξουμε και τις εξελίξεις σε ένα-δύο έτη προκειμένου αυτή η φέρπους, αν θέλετε, αποθάρρυνση των πολιτών που αντιμετωπίζουν την πολιτική πραγματικότητα την καθημερινή, να μπορέσει να τερματιστεί. Νομίζω ότι θα αποτελούσε μεγάλη ε, λειτουργία, αν θέλετε, της ομάδας μας, της Επιτροπής μας, αυτό. Ο κύριος Ντάφ ζήτησε το λόγο, γιατί ε, και μετά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πρέπει να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πρόεδρε, καταρχάς πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος το Κοινοβούλιο να παραμείνει εκτός ε, παιχνιδιού, αν θέλετε, στο θέμα αυτό. Οι, οι αλλαγές ε, που είναι απαραίτητες ε, για τη συνθήκη και που συζητώνται τώρα, προφανώς απαιτούν μία σύμβαση και το Κοινοβούλιο όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ε, συνεδρίου ή σύμβασης κτλ. είναι αρκετά ενδυναμωμένο. Εγώ θα ήθελα να προετοιμάσουμε την θέση μας πολύ προσεκτικά με δια, τις απαραίτητες διαβουλεύσεις. η γνωμοδότηση την οποία θα υποβάλουμε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων δεν είναι αυτό. Δεν είναι απλώς και μόνο μια γνωμοδότηση. Είναι σημαντικό να στείλουμε, μια... να στείλουμε κάποια σημάδια όσον αφορά τον ε, συλλογικό χαρακτήρα του Κοινοβουλίου και να ε, καταδείξουμε ότι υπάρχει συνοχή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι για να συντάξουμε μία, ένα σωστό και καλά δομημένο οικονομικό σχήμα για την διακυβέρνηση ξεπερνάει την διαβούλευση, την γνωμοδότηση αυτή και ξεπερνάει και την επιτροπή μας επί, επί του παρόντος. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εάν γινόταν κάτι τέτοιο θα πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν πιο συνενετικοί. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια διακομματική συμφωνία όσον αφορά τις θεσμικές αλλαγές που εγκρίνουμε. στην ε, ομάδα αυτή των ε, συνδέσμη των έξι οδηγιών είδαμε ποια ήταν η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποια είναι η διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση των σοσιαλιστών. Και καλό θα ήταν όντως ε, να ξέραμε ότι θα μπορούσε αυτή η επιτροπή μας να προετοιμάσει, να προετοιμάσει τον, ένα σωστό πλαίσιο για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ο Πρόεδρος, έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο για τις, που θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την ε, ψηφοφορία, ο κύριος Έφερ. Είχα ζητήσει το λόγο πριν ε, πείτε ότι θέλετε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Εν συντομία, δεν έχουμε διεξάγει τη συζήτηση αυτή στην Επιτροπή, αλλά συμφωνούμε ότι η συζήτηση δεν είναι μόνο συζήτηση για οικονομικά μέσα, τα οποία αναφέρονται στην χρηματοπιστωτική αγορά. Όχι, πρόκειται για μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια συζήτηση για το σωστό θεσμικό πλαίσιο και τη διαμόρφωσή του. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συζητηθούν και συζητιόνται. Θα ήθελα να τονίσω ότι θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το Κοινοβούλιο να παίξει ενεργά ρόλο στο σημείο αυτό. Όχι μόνο να περιμένει στα σημεία εκείνα στα οποία μπορούμε να βρούμε συνένεση θα πρέπει να καταγράψουμε τη θέση μας και να δημιουργήσουμε μια τέτοια έκθεση επισκόπησης των θέσεων αυτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους φόβους του κυρίου Ντάφ ε, για τις ε, θέσεις των διαφορετικών ομάδων και για τις ενδεχόμενα δεχασμό του Κοινοβουλίου, αυτό θα το δούμε στο τέλος αν δώσουμε εντολή για μια τέτοια έκθεση πρωτοβουλία, θα μπορέσουμε στην Επιτροπή να συζητήσουμε επί τη ουσία και θα δούμε κατά πόσον θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, σε ένα αποτέλεσμα πλειοψηφικό, ομοφωνίας. Αν δεν καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, ε, δεν θα προκύψει έκθεση. Έχουμε όσο χρόνο χρειαζόμαστε, αλλά αν δεν ξεκινήσει η συζήτηση, νομίζω ότι θα προδώσουμε κάπως την εντολή την οποία μας έχει δώσει ο κόσμος. Ήθελα να πω, λέει ο κύριος Γκολτιέρη, ότι σημειώνω ότι ο κύριος Ντάφ είναι διατεθειμένος να συνενέσει μόνο εάν προηγουμένως πούμε ότι συμφωνούμε μαζί του για το τι θα γράψουμε στην έκθεση. Δεν νομίζω ότι είναι και η καταλληλότερη μέθοδος εργασίας του Κοινοβουλίου. Πρόεδρος, προτείνω λοιπόν να ε, ξανασυζητήσουμε στο θέμα στις συνεδρία των συντονιστών. Δεν θεωρείται λήξαν το ζήτημα, παρά το γεγονός ότι το συζητήσαμε και χθε, διότι υπάρχει στο μεταξύ μία πρόταση να γίνει και μια ελεύθερη συζήτηση μεταξύ ημών για το θέμα και υπήρξαν και έντονες πιέσεις σήμερα για να συζητήσουμε το ζήτημα. Στην επόμενη συνεδρίαση λοιπόν των συντονιστών θα ξαναθέσω στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Καταρχάς έχουμε να ψηφίσουμε την έκθεση Μάρτιν. Έχετε ήδη όλες τις τροπολογίες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Άρθρο 1. Προφορική τροπολογία του κύριου Νταφ. Υπέρ. Παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομίζω σχεδόν ομόφωνα. Συμβιβαστική τροπολογία α του εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Άρθρο 1 που καλύπτεται όμως, συγγνώμη, από τη συμβαστική τροπολογία, επομένω δεν ψηφίζουμε. Συμβαστική τροπολογία B του εισηγητή, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν ε, ούτε αρνητικές ψήφιες ούτε αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η συμβαστική τροπολογία Β και Μπορούμε να θεωρούμε λοιπόν ότι καλύπτονται η τροπολογία 5. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 6 του κ. Βίλαντ. Υπέρ. Κατά. Ε, approvato. 10 contro 8. 10 contro 8. 10 ψήφοι υπέρ, 8 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 και πάλι του κ. Βίλαντ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία α, δεν ε, την ψηφίζουμε λοιπόν. Η τροπολογία 9 και πάλι του κυρίου Βίλαντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10, Βίλαντ, καλύπτεται από την συμβαστική τροπολογία Α, δεν ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 11, υπέρ παρακαλώ, του κυρίου Βίλαντ και πάλι. Κατά. Είναι. Αποχές, εγκρίνεται με μία ψήφο κατά. Φτάσαμε λοιπόν στην τροπολογία 12 Δίλαν, που έχει όμως και μία προφορική τροπολογία του εισηγητή, ο οποίος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Yeah, sorry. Ναι, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Έχουμε και πάλι το σάλ, ενώ είχαμε συμφωνήσει να βάλουμε το may, επομένως ε, witness and, Expert experts may, if this or request be heard in camera. Ναι, ναι, ναι, Μπορούμε να ψηφίσουμε, ναι, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C του εισηγητή για το άρθρο 9 παράγραφος 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. 9 a 9, quindi non, non 9 9 Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ποιο είναι υπέρ. Και Κατά. 10 ψήφοι υπέρ 8 κατά εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε τη 14 γιατί δεν πέρασε συμβαστική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Για τη 14. Κατά. non passa. 9 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 Βίλαντ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 9 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Τροπολογία 16 Ράγκελ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 Φόξ. Γλωσσική μόνο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 Φόξ, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19 Fox. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 και πάλι Fox. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία D του εισηγητή. Υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 του κύριου Φόξ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία ή όπου υπάρχει και μια, ένα αίτημα για κατατμήματα ψηφοφορίας, το οποίο όμως απορρίφθηκε. Ε, ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στην τροπολογία 22 Fox, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Φόξ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Φόξ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία F για το άρθρο 16 του εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 25 Fox. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26 Βίλαντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 Βίλαντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G. Υπέρ κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 28 Βίλαντ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 29 Βίλαντ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30 ε, την οποία υπάρχει και προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία H. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 με προφορική τροπολογία του εισηγητή της κυρίας Γιαννάκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική, ε, συγγνώμη, τροπολογία 2 Γιαννάκου, η οποία καλύπτεται όμως από τη συμβαστική τροπολογία ε που μόλις ψηφίσαμε. Τροπολογία 3 της κυρίας Γιατουνμάκη, που υπάρχει και προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. αποχέ συγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο της νομοθετικής πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως τροποποιήθηκε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν συγχαρητήρια στον κύριο Μάρτιν. Ήταν σημαντική αυτή η έκθεση, επομένως πραγματικά συγχαρητήρια κύριε Μάρτιν. Dobbiamo passare alla votazione, passiamo a questa votazione per me. Τώρα περνάμε στην ε, επόμενη στο επόμενο σημείο που είναι η ψηφοφορία για την ε, έκθεση για την ΜΕΚΙ, για την τροποποίηση του κανονισμού όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Δύο τροπολογίες έχουμε, μόνον. Και η πρώτη τροπολογία είναι καθαρά γλωσσική νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να ψηφίσουμε. Γίνεται δεκτή η πρώτη τροπολογία. Η δεύτερη τροπολογία τώρα, η τροπολογία αριθμών 1, τίθεται σε ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο κανονισμού, το σχέδιο της έκθεσης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η γνωμοδότηση και νομίζω ότι τελείωσαμε με τις ψηφοφορίες. Τώρα θα πρέπει να δώσουμε το λόγο. Νομίζω.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 Niente, posso subito dare la parola. το λόγο αμέσω. στην Αντιπρόεδρο Τζίτα Γκουρμάη που θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την έκθεση για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, η Επιτροπή ε, αναφορών είναι η καθήλυνα αρμόδια, είναι αυτή η οποία προετοιμάζει την, την έκθεση και εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Διαβάζοντα την τελευταία έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ιθαγένεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κατέστη το εξή απόλυτα σαφέ και θα σα εκπλήξει αυτό. Είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Η ηθαγένεια λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μένα σημαίνει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης ανεξάρτητα από την εθνική του προέλευση ε, έχει την ίδια, την ίδια μεταχείριση, ίδια μεταχείριση στην ίδια κατάσταση. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, τόνισε επιπλέον την ε, έννοια της ευρωπαϊκής ηθαγένειας και τα σχετικά δικαιώματα το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας κατοχυρώνονται και στον χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι νομικώς δεσμευτική. Τα δικαιώματα αυτά πέρα από το ότι ορίζονται στο πρωτογενές δίκαιο αναπτύσσονται και στο δευτερογενές δίκαιο. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των ε, κανόνων και τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά διασυνοριακές καταστάσεις και όλοι το ζούμε αυτό. Στο χαρτί όλα φαίνονται όλα πολύ ωραία, αλλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και στην πράξη. Αυτό δεν είναι απλό. Πώς θα καταστεί λοιπόν δυνατόν για 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να νιώσουν πραγματικά στην καθημερινότητά τους τα ωφέλη της ευρωπαϊκής ε, ηθαγένειας. Συνάδελφοι, όταν κατέρτισα την ε, γνωμοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη και της αρμοδιότητας της Επιτροπής μας, πρότεινα μια διτή προσέγγιση. Καταρχάς, οι πολίτες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση σε ό,τι αφορά τα εκλογικά τους δικαιώματα. Θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση και να θέλουν επίσης να συμμετέχουν. Δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε φυσικά να συμμετάσχουν. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί μια ιστορική ανάγκη τους. Είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να προκαλέσουμε αυτό το ενδιαφέρον και αυτή την προσέγγιση ακολουθώ και ακολουθούν οι πιο πολλές από τις προτάσεις μου. Μιλώντας λοιπόν για την ε, ενημέρωση. Θα πρέπει να καλύψουμε πολλούς τομείς. Χρειάζεται σωστή και κατανοητή ενημέρωση από μια σειρά πηγών από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από τα κράτη-μέλη. Σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρξει ερμηνεία, ανάλυση και ενημέρωση των πολιτών. Και εδώ λοιπόν εμείς οι πολιτικοί αλλά και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα πρέπει να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο. Ενημέρωση μπορεί να σημαίνει εκστρατείες ε, ενημερωτικές όπως για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το έτος 2013 ως το έτος του Ευρωπαίου Πολίτη. Και ασφαλώς θα αποτελέσει και το επόμενο έτος των ευρωπαϊκών ε, των ευρωεκλογών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτή η πληροφόρηση, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά σημαντικά και σπουδαία ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να προβληθούν καλύτερα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή. Είναι σημαντικό το δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών και αυτή η συμμετοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από πολλές μορφές. Το πιο σημαντικό είναι η συμμετοχή στις εκλογές, είτε σε ό,τι αφορά το εκλέγην, είτε σε ό,τι αφορά το εκλέγεστε. Να σας υπενθυμίσω ότι 42% των πολιτών προσήλθαν στις κάλπες το 2009. Λίγος κόσμος πηγαίνει στις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτομα που ζουν εκτός της χώρας τους. Χαίρομαι που το έθεσες αυτό στη γραπτή σου ερώτηση, Άντριου, σε ό,τι αφορά την συνέχεια τους διαδόχους, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι χρειάζονται δυνατά, δυναμικά ευρωπαϊκά σύμβολα για να αυξηθεί η συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Μιλώντας για θέματα συμμετοχής, είμαι βέβαιη ότι όλοι θα περιμένετε να αναφέρω το νέο νόμο της συνθήκης της Λισαβόνας. Όλοι φυσικά ξέρετε την Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία των Πολιτών που θα ισχύσει σύντομα. Οι συγητές λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει το έργο μας, αλλά νομίζω ότι πλέον επαφίεται, αναπόκειται στα κρατημέλη να εφαρμόσουν όλους τους νόμους προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να συμμετάσχουν πιο ε, εντατικά στην καθημερινή ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι την εφαρμογή ε, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για να επεκτείνουμε το δημοκρατικό αυτό εργαλείο. Εν συντομία λοιπόν αυτά τα σχόλιά μου και ασφαλώς θα χαρώ να διαβάσω και τις δικές σας ιδέες. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την συνάδελφό μας, την κυρία Γκουρμάη, και αυτή την τόσο εμπνευσμένη γνωμοδότηση, την φιλική προς, το, προς τους πολίτες. Αυτό δεν θα έπρεπε να μας ε, εκπλήξει βέβαια από αυτήν. Είναι ένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, το οποίο κάνει τις σωστές διαπιστώσεις και θέτει τις σωστές ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου, μια και αναφέρουμε την πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και τον ρόλο που έπαιξε η συγκήτριά μας για την ε, δημιουργία αυτής της πρωτοβουλίας, θα ήθελα να αναφερθώ και στον άλλο εισηγητή, στον Αλέαν Λαμασούρ, που ήδη από το 2008 είχε υποβάλει στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Ιούνιο του 2008 συγκεκριμένα, μια πλήρη έκθεση για τα δικαιώματα των πολιτών στην Ευρώπη. Μια έκθεση η οποία έκανε μια πλήρη ανάλυση, μια λεπτομερή ανάλυση όλων των εμποδίων, όλων των δυσλειτουργιών, όλων των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι ευρωπαϊκοί πολίτες ε, όταν ήθελαν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Ήταν μια έκθεση η οποία προέβλεπε, αν θέλετε, πολλά πράγματα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά από τα μέλη της Επιτροπής μας για το θέμα αυτό και θα πρέπει να διαπιστώσουμε, όπως και η συγκητριά μας βέβαια, ότι η, ευρωπαϊκή ηθαγένεια δεν ε, ε, εμπνέει, αν θέλετε, ένα αίσθημα ε, στους πολίτες ότι ανήκουν σε μια ενότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι λειτουργεί έξω από αυτούς, δίπλα από αυτούς. Ε, παρά τα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε επίπεδο επιτροπών, στην δικιά μας επιτροπή, είτε ε, σε, για, τα, για άλλα θέματα, όπως είχε προτείνει και ο Επίτροπος Μπαγνιέ, ε, μια σειρά μέτρων για την απόκτηση περισσότερης εμπιστοσύνης στην εσωτερική αγορά. Λοιπόν, όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται εδώ και σε όλα τα επίπεδα, επίσης βοηθούν. Θα ήθελα, εκτός από τα δικαιώματά μας, σαν Ευρωπαίοι πολίτες, θα πρέπει να διευκρινίσουμε καταρχάς ε, μέσω μιας καλύτερης ε, κοινοποίησης ε, να ξέρουν οι πολίτες ποια είναι τα δικαιώματα τα και συμφωνώ εδώ με την ε, ε, εισηγήτρια ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία ημερομηνία για τις ευρωπαϊκές εκλογές ή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα το οποίο θα μπορούσε να ενδυναμώσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ε, ηθαγένειας του Ευρωπαίου πολίτη. Επίσης θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο των Ευρωπαϊκών ευρωπαϊκών κομμάτων των, ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. Είχαμε την ευκαιρία να συντάξουμε και μία έκθεση για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να συνεχιστεί το έργο ε, των ε, ευρωπαϊκών κομμάτων και των Ινστιτούτων, γιατί μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην, ε, στο, στο αίσθημα του, της ευρωπαϊκής ηθαγένειας γιατί τα κόμματα ε, είναι πιο κοντά στους πολίτες. Επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στις ε, αρμοδιότητες και στα ε, και στις δυνατότητες που έχουν τα πολιτικά κόμματα. Άρα θα πρέπει να παρακολουθούμε και τι γίνεται, αν θέλετε, σε επίπεδο ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ε, όσον αφορά την ε, ε, εκπαίδευση και την, την ενημέρωση των στελεχών τους που έχουν να παίξουν έναν ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών. Επίσης, θα πρέπει και στα κράτη-μέλη να τονίσουμε την ανάγκη να περάσουν σε δράση έτσι ώστε αυτές οι πρωτοβουλίες για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια να εφαρμοστούν την άνοιξη της επόμενης χρονιάς, όπως όλοι ελπίζουμε. Θα ήθελα επίσης να κάνω ένα μικρό σχόλιο για ένα από τα θέματα τα οποία θίγει η συγκητρία στο σχέδιο γνωμοδότησης και αφορά το γεγονός ότι όλοι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν δικαίωμα στις περιφερειακές ε, ε, ε, εκλογές στα κράτη όπου οι περιφέρειες ασκούν νομοθετική εξουσία. Εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ προσεκτικά γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο πρόωρο αυτή τη στιγμή να διευρύνουμε το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές όλων των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Το να συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι ήδη μια πρόκληση. Το να, τους, ε, ε, να επιτρέπουμε στους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν σε μια άλλη χώρα εκτός από τη δική τους να συμμετέχουν σε περιφερειακές εκλογές ή σε δημοτικές εκλογές, ε, γιατί τις δημοτικές έχουν το δικαίωμα, είναι μια τεράστια πρόκληση και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι μια η διαφωνία μου. Επίσης, ε, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε, να βρούμε τρόπους για να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες μας, γιατί όλοι έχουμε αυτή την ευθύνη να ενημερώσουμε, ε, να εκπαιδεύσουμε, θα θέλετε, τους, πολι... τους πολίτες μας. Οι... βουλευτές, Ευρωπαίοι βουλευτές είναι πιο δραστήριοι και αυτοί ε, μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. θα πρέπει στα μέσα να προωθούμε τον ρόλο των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και πιο συγκεκριμένα και τον ρόλο και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες για το καθημερινό έργο το οποίο ε, εκτελείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει με τον τρόπο αυτό πιστεύω ε, να κάνουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να ενδιαφερθούν περισσότερο ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμμετέχουν ε, αν θέλετε στα τεκτενόμενα και με τον τρόπο αυτό να αποκτήσουν μια πολύ πιο δυνατή, ένα πιο, πιο, πιο δυνατό αίσθημα ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Αυτά τέλος πάντων. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε και έναν ένα ρόλο για μας στα μέσα μεζικής ενημέρωσης σκέφτομαι και, τους, και την νεολαία που συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα, πρόγραμμα Λεωνάρντο κτλ, που εποφελούνται από την ε, κοινοτική χρηματοδότηση ε, και σε επαγγελματικό και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να καλυφθεί ένα κενό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους βοηθάει πάρα πολύ, τους δίνει χρήματα, ε, εποφελούνται από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν το γνωρίζουν. Η γνώση τους όσον αφορά την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, παρουσιάζει κενά. Επομένως πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και από τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν ένα είδος μαθήματος αγωγής του πολίτου, του Ευρωπαίου, μιας αγωγή, ενό μαθήματος αγωγής ενός Ευρωπαίου πολίτη. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί βέβαια σε αυτό το θέμα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει και τα παιδιά και οι νέοι να εκπαιδεύονται και στην, και στην αγωγή του Ευρωπαίου πολίτη. Ήδη υπάρχει το, το μάθημα πολιτικής αγωγής. Ε, θα πρέπει να μην ε, παραμείνουμε βέβαια ε, μόνο στην επίσημη ιστορία, αλλά θα πρέπει, αν θέλετε, κάπως ε, να αγγίξουμε, να μπορέσουμε να αγγίξουμε και τα παιδιά. Γιατί αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, η αγωγή ενός Ευρωπαίου πολίτη. Δεν θέλω να μακρηγορήσω υπερβολικά, ε, γι' αυτό σταματάω εδώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την τόσο πλήρη παρέμβασή σας. Ο κύριος Ντάφη ζητάει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκουρμάη για τη γνωμοδότησή της. Είναι μεγάλη. Νόμιζα ότι υπήρχε κάποιος περιορισμός για τις γνωμοδοτήσεις. Αυτό το μήκος είναι μεγάλο μάλλον. Όπως γνωρίζετε δεν είμαι και υπέρμαχος της ιδέας της ε, ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Μάλλον με τρομάζει η ιδέα του Ευρωπαϊκού Δήμου και μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην παράγραφο 4. Θα ήθελα να επισημάνω παρόλα αυτά ότι η δεύτερη εκθεσή μου για την εκλογική μεταρρύθμιση συζητάτε και ολοκληρώνεται η συζήτηση στην Επιτροπή και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο συνεπείς ε, στα όσα λέμε για τις εκλογές. Και στη γνωμοδότηση αυτή και στην έκθεσή μου. Για παράδειγμα, στην παράγραφο 9 δεν είμαι βέβαιος ότι το σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αποτρέψει τους πολίτες από το να ψηφίσουν. Νομίζω ότι είναι το αντίθετο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον κόσμο να ψηφίσει. Δεν, ε, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω κατά πόσον έχουν την ενέργεια να ψηφίσουν ε, δύο φορές ή όχι. Αυτό είναι θέμα συνείδησης. Και για μας δεν είναι κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα αυτό. Επίσης, μου είναι δύσκολο να κατανοήσω και την παράγραφο 6, η οποία η, στην αγγλική της εκδοχή τουλάχιστον λέει ότι ε, αναλογικά λιγότεροι πολίτες εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους για να ψηφίσουν. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κυρία Γκουρμπάιν τι εννοείτε. θέμα του να μην ε, αναφέρονται οι πολίτες για τις εκλογές στα Εθνικά Κοινοβούλια, που είναι και θέμα μιας προφορικής ερώτησής μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα πρέπει να συγχαίρεται με την ποιότητα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Αναρωτιούνται οι πολίτες τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει να μην μπορούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές. Και παρά το γεγονός ότι το θέμα αυτό είναι εκτός πεδίου της συνθήκης, νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα μας ανοίξει νέους δρόμους για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Apart from that, um, Πέραν αυτού όμως νομίζω ότι είναι καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέφνερ. Äh, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και ιδιαίτερα την Ζηταγκούρμα για την νομοδότηση αυτή την οποία θεωρώ ότι επί της αρχής ε, είναι καλή και με βρίσκει σύμφωνο και νομίζω ότι περιλαμβάνει και τα σημαντικά στοιχεία α, της έκθεσης. Θα είμαι σύντομος, επειδή δεν έχω άλλωστε και πολλά να προσθέσω. Μία ερώτηση μόνο θα ήθελα να ε, διευκρινίσω κάπως καλύτερα, ε, επειδή δικαίως μιλάτε ότι άτομα τα οποία προέρχονται από ένα κράτος μέλος και βρίσκονται και ζουν σε ένα άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ε, τοπικές εκλογές. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στις εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι επί της αρχής σε ό,τι αφορά της ευρωπαϊκές, την ευρωπαϊκή ηθαγένεια δεν είναι αποδεκτή η πραγματικότητα να βρίσκεται και να μετακομίζει κάποιος από μια χώρα σε άλλη και να αφήνει τα εκλογικά του δικαιώματα στην ε, χώρα του. Νομίζω λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάτσουμε και να συμφωνήσουμε, να ορίσουμε ένα χρονικό πλαίσιο με το οποίο ένας πολίτης θα μπορεί να ε, έχει δικαίωμα να ψηφίζει στην καινούργια του χώρα. Ξέρω ότι θα προκληθεί σύγκρουση με το εθνικό δίκαιο δεν είναι απαραίτητο αυτό να γίνει στα πλαίσια της παρούσας γνωμοδότησης, αλλά θα πρέπει να το λάβουμε στα σοβαρά αυτό, γιατί το δικαίωμα του εκλέγει να αποτελεί το κατεξοχήν δικαίωμα του πολίτη για την διαμόρφωση του πολιτικού γίγνεσθε. Και το γεγονός ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να γίνει αξιοποίηση του δικαιώματος αυτού θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το βιώσιμο. Δεν θα πρέπει να κλείνουμε επίσης τα μάτια και να αγνοούμε τις πολλές ε, εξελίξεις, τις σωτικές εξελίξεις, την μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ενημέρωση. Αλλά μιλώντας για θέματα ηθαγένειας δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι η εμπιστοσύνη των ε, πολιτών στα θεσμικά όργανα φθήνει και πάει. Υποχωρεί. Ιδιαίτερα με τις τρέχουσες εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές. Δεν πρόκειται να πετύχουμε κάποια βελτίωση της κατάστασης. Δεν πρόκειται να καταφέρουμε να δώσουμε την αίσθηση στους πολίτες ότι εκπροσωπούμε τα συμφέροντά τους και ότι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της κατάστασης. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην εκκίνηση, στην πρώτη της φάση και δεν έχουμε σε καμία περίπτωση ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Είπατε επίσης και συμφωνώ απόλυτα ότι είναι σημαντική η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να καταστεί επιτυχής αυτή η πρωτοβουλία και νομίζω ότι αυτό θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων και από τις υποδομές που θα αναπτυχθούν για την πρωτοβουλία αυτή και από πολλά άλλα στοιχεία. Άρα είναι και δική μας ευθύνη να καταστεί επιτυχής αυτή η πρωτοβουλία και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χέφνερ, κύριο Σέπφλιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας ξεκινήσω επιστήοντας, επι, ε, υπογραμμίζοντας την παράγραφο 6. Έχετε δίκιο εδώ σε αυτό που λέτε, όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Διότι και αυτό ισχύει για όλα τα νομοθετικά κείμενα. Πιστεύω ότι εδώ ξεπερνάμε απλώς το ερώτημα τι κάνει, τι δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε πολλούς παράγοντες, νέους παράγοντες. Έχουμε την κοινωνία των πολιτών, υπάρχει η παγκοσμιοποίηση, εκεί δεν υπάρχει σε, σε ορισμένους τομείς πολιτικός έλεγχος. Επομένως όλοι οι νομοθέτες αντιμετωπίζουν ένα ανάλογο πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν σχολιάζουμε τους ψηφοφόρους που δεν συμμετέχουν ε, στις ευρωπαϊκές εκλογές. Όντως, η συμμετοχή στις εκλογές είναι χαμηλή. Μία παρατήρηση αυτή. Δεύτερη παρατήρηση, παράγραφος 10. Δεν είναι σαφές για μένα τουλάχιστον τι σημαίνει εδώ περιφέρειες που έχουν νομοθετικές αρμοδιότητες. Μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, για κάτι διαφορετικό από την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλό θα είναι να το διευκρινίσουμε αυτό. Τρίτο σημείο, παράγραφοι 7 και ως 11. Για τους συμβολισμούς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι οι συμβολισμοί είναι σημαντική σε όλο το πολιτικό σύστημα και όσοι το αρνούνται ε, έχουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα για το, τα όσα γίνονται. Όμως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν σύμβολα, μπορεί να μην έχουν ενταχθεί άμεσα στο, στη συνείδηση των πολιτών, αλλά όταν, ας πούμε, οι πολίτες, σε αποτέλεσμα όμως, οι πολίτες δεν μπορούν να αναγνωρίσουμε ένα τον άλλον. Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε την πολιτική πραγματικότητα ότι τα κράτη είναι αυτά που κάνουν που ορίζουν την καθημερινή ζωή. Ναι, μεν έχει αναλάβει, έχει εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σημαντικό μερίδιο εξουσίας, όμως την βασική εξουσία την ασκούν τα κράτη-μέλη, αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την αγνοούμε. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να διατυπώσουμε τροπολογίες για αυτά τα θέματα, αλλά είναι σημαντικό να τα εκφράσουμε. Είναι ότι το 98% και εδώ είμαι γενναιόδωρος, είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουν ε, ότι, υπάρχουν, ε, ότι έχουν μάλλον μια διπλή ταυτότητα ως, ως πολίτες. Δηλαδή ότι είναι πολίτες της χώρας τους, αλλά και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το διτό, αν θέλετε, το δυσυπόστατο, δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν εύκολα. Θα μπορούσε να γίνει ε, μια συγκεκριμένη έκθεση για, το, για, το, για αυτό το θέμα θυμηθείτε τι έγινε με το Ιρλανδικό δημοψήφισμα που είχαν αποσυνδεθεί εκεί. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ε, ότι ήταν πολίτες και των δύο οντοτήτων τέλος πάντων. Η πολιτική ελίτ, η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη είναι και αυτή διαιρεμένη ε, ανάμεσα στην εγχώρια πολιτική τάξη και σε μας. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο για να καλύψουμε αυτό το κενό. Εδώ τώρα. Εδώ αυτή η αύξηση της διακυβερνητικής, ε, των διακυβερνητικής αρμοδιότητας πιστεύω ότι δεν βοηθάει. Είμαστε στο 0-0 εδώ, πιστεύω. Δηλαδή δεν, δεν ε, βοηθάει σε τίποτα. Τώρα για την ε, παράγραφο 11 που αναφερόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεωρηθεί ένα παράγοντα στην εσωτερική πολιτική ζωή των κρατών μελών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μένα, αλλά θα προκαλέσει και αντιδράσεις και στους ευρωσκεπτικιστές, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν καλές προθέσεις. Γιατί δεν μπορούν ε, να δουν ε, ποια είναι η σχέση, αν θέλετε, τι δουλειά έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό των κρατών μελών. Λοιπόν, η ιδέα ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, είναι άμεση παράγοντες ε, ρύθμισης ε, της εσωτερικής πολιτικής ζωής των κρατών μελών είναι κάτι που αυτή τη στιγμή το θεωρώ ιδιαίτερα πρόωρο και δεν, και δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε όμως, πιστεύω, ότι θα μπορούσαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να ελέγξουν τον τρόπο εφαρμογής και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη, που διαφέρει από κράτος σε κράτος, σε κράτος μέρος. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που δεν το έχουμε λύσει αυτή τη στιγμή. Εγώ στην Ουγγαρία το αντιμετώπισα αυτό το πρόβλημα με τους ε, ε, ψηφοφόρους μου Α, και κάτι άλλο τώρα, μια παρατήρηση για τον Άντριου, στον Άντριου Ντάφ. Αυτό το οποίο έχουμε εδώ η, η Ευρώπη από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον δεν, δεν έχει απομακρυνθεί πολύ από την εικόνα που είχαμε πριν από 50 χρόνια. Δεν υπάρχει πολιτική συνείδηση όμως πιστεύω. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκοί δήμοι, αν θέλω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ευρωπαϊκό δήμο. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και το και Eurovision. Εκεί όντως η Ευρώπη ενώνεται. Πρόεδρος, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, άλλες παρεμβάσεις. Ε, η συγγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που τόσοι συνάδελφοι πήραν το λόγο και κατέθεσαν τροπολογίες για να σχολιάσουν ήταν πολύ καλή η εισήγησή σας. Δεν θα ήθελα να ανοίξω το κουτί της Παντόρας, αλλά ασφαλώς και χρειάζεται μια τέτοια συζήτηση εδώ στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα σχόλιά σας. Ασφαλώς όλα τα σημεία τα οποία θίξατε είναι έγκυρα. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρετε να καταθέσετε τέτοιες τροπολογίες. Ξέρω ότι δεν είναι απλό το εγχείρημα στη συγκεκριμένη περίπτωση και ο συνάδελφος κ. Σόπφλινγκ ξεκαθάρισε ότι ασφαλώς αυτό δεν αποτελεί κάτι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ασφαλώς. Δεν ήταν εύκολο να κατακτηστεί και η έκθεση και η γνωμοδότηση και μας πήρε και κάποιο χρόνο. Θα ήθελα όμως να ενδυναμώσετε και να εμπλουτίσετε τη θέση μας και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την τελική μας τοποθέτηση. Και ασφαλώς, επειδή προερχόμαστε και από διαφορετικό πολιτισμικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, είναι διαφορετική και η προσέγγιση μας σε ό,τι αφορά τις τοπικές εκλογές. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε και το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ που αναφέρατε την επόμενη γενιά. Γιατί ποιος θα αναλάβει στο μέλλον το έργο μας αν δεν εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά. Και προς το παρόν η επόμενη γενιά μας στήσεται από ανεργία. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να μας απασχολήσουν σε ό,τι αφορά τα σχολεία. Πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα γιατί θα πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε, ανήκουμε στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης το θέμα της εθνικής ή της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Νομίζω ότι και οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να συνδράμουν στο σημείο αυτό, γιατί αν τώρα μιλάνε, αν κάποιος μιλάει με διπλή, διτή ιδιότητα και λέει ότι αν τώρα μιλώ υπό την ιδιότητά μου ως εθνικός πολιτικός ή ως ευρωπαϊκός πολιτικός, όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τους Βρυξέλλες ενθαρρύνονται. Και γι' αυτό εν μέρη αυξάνεται αυτός ο εξτρεμισμός στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει και κάποια ευθύνη των πολιτικών ηγετών. Και συμφωνώ επίσης σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της ψήφου. Θα πρέπει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο να αναλογιστούμε τέτοια ζητήματα. Θεωρούμε ασφαλώς ότι είναι θαυμαστό εργαλείο η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, αλλά δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τελικά. Συναντήθηκα και με την ομάδα επικοινωνίας του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με ρώτησαν τι θα συμβεί αν το Συμβούλιο αν τα κρατημέλη δεν είναι έτοιμα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι θέμα που μπορώ να απαντήσω εγώ, αλλά δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να απευθύνουμε ένα σαφές αίτημα προς την Προεδρία για να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η κατάσταση, τι γίνεται με το ECI, με αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό τώρα Δήμο, το Ευρωπαϊκό Εκλογικό Κοινό. Φυσικά υπάρχει, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ταυτότητες σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά κατά την ε, ψηφοφορία. Φυσικά διαφέρουν τα πράγματα στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές. οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν αυτό που επιθυμούν. Και μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δεν νομίζω ότι συμφέρει κανέναν να παραμελήσουμε τα θέματα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία θα παίξει σημαντικό ρόλο για την επανασύνδεση των πολιτών. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω λοιπόν να καταθέσετε καλές τροπολογίες σε ό,τι αφορά τώρα το μέγεθος του κειμένου. Δεν ξεπέρασα τις προδιαγραφές και κατά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία έμαθα ότι είναι καλό να είναι συνεκτικό ένα κείμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να περιορίσουμε το κείμενο, να μου πείτε ποιο ε, κομμάτι θεωρείτε ότι είναι περιττό, ότι θα μπορούσαμε να το αφήσουμε έξω. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα σχόλιά σας συνάδελφοι. Θα χαρώ να λάβω τις τροπολογίες σας. Να σας πω ότι πήρα πολύ στα σοβαρά την ε, δουλειά. Μπορούσα να αποφασίσω να εργαστούμε μόνο με την αγγλική εκδοχή του κειμένου επέλεξα να έχουν όλοι οι συνάδελφοι την γλώσσα τους με τη βοήθεια της γραμματείας. Νομίζω ότι και αυτό αποτέλεσε έκφρασε του σεβασμού μου προς τους συναδέλφους για να δουλεύει ο καθένας με τη γλώσσα του. Ελπίζω λοιπόν να είναι τελικά καλή η γνωμοδότηση και να λάβει την υποστήριξη όλων των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι αυτή που ζήτησε την γνωμοδότηση, θα πρέπει να υιοθετήσει στις 22 Νοεμβρίου την έκθεση αυτή, θα μπορούσαμε να ε, ορίσουμε ημερομηνία προθεσμία για την υποβολή των ανατροπολογιών μας 27 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Πολύ ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η έκθεση του κυρίου Μέσσερ για την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί το καθεστώς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε καθυστερήσει λίγο, διότι η νομική επιτροπή που είναι υπεύθυνη θέλησε να περιμένει την γνωμοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την έχουμε στη διάθεσή μας. Και δίνω αμέσως το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μέσσερ Σμιτ. Thank you, Chair. Um, yes, I can. Πρόεδρε, να σας επιβεβαιώσω λοιπόν αυτά που είπατε. Περιμέναμε τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα επειδή την έχουμε θα μπορέσουμε να τη συμπεριλάβουμε στην έκθεση και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Το ιστορικό βέβαια είναι η πρόταση του δικαστηρίου να αναδιοργανωθεί λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στο φόρτο εργασίας τα τελευταία 10 χρόνια, από το 2000 έως το 2010 είχαμε μια αύξηση της τάξης του 65% των δικαστικών υποθέσεων, το οποίο είναι ανάλογο με αυτό που έχουμε και στα άλλα διεθνή δικαστήρια και στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, που είχαμε αντίστοιχη αύξηση του φόρτου εργασίας και αυτό οδήγησε σε θεσμικές αλλαγές και σε αυτό που διαπιστώνουμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο είναι ότι οι δικαστές παρουσίασαν τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του έργου τους, διασφαλίζοντας ε, ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις ε, στο δικαστήριο δεν θα καθυστερήσουν, θα τηρούνται και υποχρεώσεις για το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη ε, και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ε, συντομία λοιπόν να πω τις τέσσερις προτάσεις στα του δικαστηρίου, στα μέλη της Επιτροπής και το τι προτείνω εμείς να γράφουμε στη γνωμοδότηση για τις προτάσεις του δικαστηρίου. Καταρχάς, το δικαστήριο προτείνει να υπάρχει ένα γραφείο αντιπροέδρου του δικαστηρίου και να εφαρμόσει τα όσα κάνουν οι αντιπρόεδροι στο έργο του δικαστηρίου. Δηλαδή, οι αρμοδιότητες του Προεδρού, επειδή ακριβώς αυξήθηκε ο φόρτος εργασίας, ε, θα παρακολουθούνται ε, πιο επισταμένα από τους αντιπροέδρους. Δηλαδή, θα είναι πολύ πιο στενή συνεργασία αντιπροέδρων και προέδρου. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι λογική αλλαγή. Γι' αυτό ακριβώς πρότεινα να είμαστε υπέρ αυτής της αλλαγής. Η δεύτερη πρόταση στη σύνθεση του δικαστηρίου αφορά τον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργεί η, το δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 δικαστές και προτείνεται να αυξηθεί ε, στους 15 δικαστές για να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα ε, που υπάρχουν με την αύξηση του φόρτου εργασία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπέρ και αυτή τη αλλαγή. Μία από τις πιο διαφιλονεκούμενε προτάσεις είναι η δυνατότητα να υπάρχουν και αναπληρωτές δικαστές ε, στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Προτείνεται κάποιοι από αυτούς τους δικαστές ε, οι οποίοι έχουν αποσυρθεί να συμπεριλαμβάνονται σε ένα κατάλογο και σε περίπτωση που οι τακτικοί δικαστές πρέπει να απουσιάσουν για τρεις μήνες για, τουλάχιστον λόγω ε, ιατρικών θεμάτων, να μπορούν αυτοί οι αναπληρωτέ δικαστές να τους αντικαταστήσουν. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα για δύο λόγους τουλάχιστον. Καταρχάς, οι δικαστές αυτοί ε, κατά βάση θα μπορούν να συμμετάσχουν στο δικαστικό έργο και όχι, μόνο στα, και όχι στα διοικητικά καθήκοντα, τα οποία είναι και αρμοδιότητα των δικαστών ε, ε, εν το μέσο των δικαστικών υποθέσεων και κατά την άποψή μου θα δημιουργήσει και μία ε, κατηγορία ε, δεύτερης υποστάθμης δικαστών που νομίζω ότι δεν είναι προς το συμφέρον των δικαστηρίου η εσωτερική ισορροπία μεταξύ των δικαστών μπορεί να διατηρηθεί και φυσικά μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα κατά την ε, έκδοση των αποφάσεων. Τα μέρη που έχουν λάβει μία απόφαση από το δικαστήριο, πώς μπορεί να νιώθουν ε, όταν υπάρχει μία σύνθεση στην οποία συμμετείχαν αυτοί οι αναπληρωτές δικαστές ε, και να νιώθουν ότι είναι μία απόφαση της ίδιας αξίας η οποία ε, με μία απόφαση που έχουμε λάβει από τους μόνιμους δικαστές. Νομίζω ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα εδώ. Γι' αυτό ακριβώ και ζητώ από τα μέλη της Επιτροπής να μου πούν την άποψή τους ε, για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί έχω αμφιβολίες για το κατά πόσον πρόκειται για σωστή πρόταση και σωστό τρόπο αντιμετώπιση από το δικαστήριο. Ίσως θα έπρεπε εδώ να ακούσουμε και την άποψη των μελών. Η τέταρτη και τελευταία σημαντική πρόταση αλλαγής είναι μια πρόταση για το Γενικό Δικαστήριο που προτείνεται να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών από τους 27 που έχουμε σήμερα στους 39, να προσθεθούν δηλαδή 12 μέλη. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται να υπάρχουν πιο εξειδικευμένα δικαστήρια. Όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δικαστήριο πιο εξειδικευμένης φύσεως, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, αλλά προτείνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο να απορρίψει την αύξηση των αριθμών, του αριθμού των δικαστών ένας τρόπος αντιμετώπισης ε, της αύξησης του φόρτου εργασίας, ε, όπως προτείνεται εδώ, είναι να υπάρχουν πιο εξειδικευμένα δικαστήρια. Για παράδειγμα, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται από το ε, νέο ειδικό δικαστήριο. Όλα αυτά προκύπτουν από ανάγκη για πιο αποτελεσματική λειτουργία του δικαστηρίου και μεγαλύτερη ευελιξία. Εδώ έχουμε δύο εναλλακτικέ λύσεις. Είτε να αυξηθεί ο αριθμό των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο ή να υπάρχουν περισσότερα ειδικά υποδικαστήρια, αν θέλετε. Κατ' εμέ, ο καλύτερος τρόπος να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο ευέλικτοι τις εργασίες μας, ιδίως όσον αφορά τις υποθέσεις εν εξελίξη είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστών και όχι να αρχίσουμε να συστήνουμε ε, ειδικά δικαστήρια σε πιο εξειδικευμένους τομείς. Η πρότασή μου, αφού είδα και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι να ε, αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστών κατά 12, όπως προτείνεται στο δικαστήριο. Έχουμε και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, επισυνάπτεται στο φάκελό σας. Για την πρώτη πρόταση, για τη δημιουργία ε, γραφείου αντιπροέδρων, εδώ έχουμε ε, την ίδια άποψη με τη δική μου, θα μπορούσαμε να δεχτούμε δηλαδή την πρόταση αυτή. Όσον αφορά τώρα την ε, τροποποίηση του αριθμού των δικαστέων από 13 σε 15 στο τμήμα μείζωνος συνθέσεως ε, λέγεται ότι και αυτό είναι λογικό γιατί μπορούμε έτσι να αντιμετωπίσουμε την αύξηση του φόρτου εργασίας. Όσον αφορά τώρα τους ε, προσωρινούς δικαστές, τους αναπληρωτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να είναι υπέρ της θέσης του δικαστηρίου και αυτό πρέπει κάπω να αντικατοπτρίζεται και στη γνωμοδότησή μας. Δεν θεωρώ όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξετάζει καμία από τις ανησυχίες που έχουμε εμείς, το να έχουμε δηλαδή δεύτερης κατηγορίας δικαστές ε, στο δικαστήριο και νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να το εξετάσουμε, όχι μόνο όσον αφορά τα εσωτερικά ζητήματα και την εσωτερική κατανομή του έργου του δικαστηρίου, αλλά κυρίως ε, όσον αφορά τους διαδίκους που θα πρέπει να δεχτούν την απόφαση του δικαστηρίου και πώς θα νιώθουν αν ένα ή δύο από τους δικαστές που ε, εξέδωσαν απόφαση για την υπόθεσή τους είναι αναπληρωτές δικαστές. The fourth ε, question where we have to choose either to... Και για το τέταρτο θα πρέπει να αποφασίσουμε ή αύξηση του αριθμού των δικαστών ή να έχουμε περισσότερα ειδικά δικαστήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή θεωρεί ότι το θέμα είναι επίγον και πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι, είναι υπέρ της αύξησης του αριθμού των δικαστών, όπως προτείνω και εγώ. Αυτά τα τέσσερα ζητήματα λοιπόν είναι και η προτάση του δικαστηρίου. Κατόπιν, έχω προσθέσει και ένα πέμπτο σημείο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό ε, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, είμαστε σε μια ε, χρονική στιγμή όπου όλοι ζητούν να είμαστε πιο ευέλικτοι, πιο ελαστικοί και βλέπουμε ότι και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο ε, στο μέλλον λόγω της προσχώρησης της σύμβασης ε, και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πιο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί διαπιστώνουμε ότι ακολουθείται αυτή η διαφάνεια και ο πιο ανοιχτός χαρακτήρας και επιτρέπουν και αποκλίνουσες απόψεις ε, στο δικαστήριο, την αποκλίνουσα γνώμη και νομίζω ότι το ίδιο θα πρέπει να έχουμε και εμείς. Όπως ε, δουλεύει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ίδιο να επιτρέπεται και για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να εκφράζεται η άποψη της μειοψηφίας σε κάποιες περιπτώσεις και νομίζω ότι αυτό συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές της συνθήκης της Λισαβόνας και τουλάχιστον θα δώσει και τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα και να εφαρμόζονται σωστότερα ε, οι διάφορες πτυχές, διότι έτσι η πλειονότητα των δικαστών θα μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους για την έκδοση μιας συγκεκριμένη απόφασης και ταυτόχρονα να διασκεδάσουν και τις αμφιβολίες που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιες αποφάσεις. Είδαμε ότι υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα επιθελούσες βάσεως στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο θα έπρεπε εμείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να είμαστε λιγότερο ανοιχτή και διάφανη ε, για τους πολίτες αλλά και για όσους εργάζονται στο δικαστήριο και εκτός δικαστηρίου από ότι το δικαστήριο στο Στρασβούργο. Ολοκληρώνω λοιπόν και θα σας δώσω τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα. Ε, να πω ότι οι δικαστές θα αποφασίζουν ε, μόνο εάν θα θέλουν να εκφράζεται και η αποκλίνουσα γνώμη στις αποφάσεις, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε το ίδιο ανοιχτοί στο δικαστικό σύστημα όπως ε, θέλουμε να είναι και η πολιτική μας ε, και όλοι οι υπόλοιποι. Πολλές φορές σας έχω αποστείλει τις προτάσεις μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μου απάντησαν και είναι διατεθειμένοι να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Προσβλέπω λοιπόν στη συζήτηση και Έχω αποστείλει και την άποψή μου για αυτή την αποκλίνουσα γνώμη στο δικαστήριο και η απάντηση που έλεγα ήταν ότι θεωρείται ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε, για το οποίο συγγνώμη, θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς οι πολιτικοί και δεν θα πρέπει ε, να λάβουν κάποια θέση ε, επί του ζητήματος δημοσίως. Το σεβόμαστε αυτό αλλά ελπίζω να συνεισφέρετε και εσείς με τις απόψεις σας ε, για την έκθεση αυτή. Το σχέδιο κειμένου είναι στη διάθεσή σας και είμαι και εγώ στη διάθεσή σας για προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μέσσερ Σμίτ. Γουαλτιέρη, Νταφ και Έφνερ είναι αυτοί που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Γκουαλτιέρη. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, εργασία που έκανε και γιατί ακριβώς ε, συνέλαβε το πνεύμα της συνθήκης. Γιατί εδώ, για αυτού του είδους των μεταρρυθμίσεων, της μεταρρυθμίσης, προβλέπεται η συναπόφαση και δεν περιορίζει το ρόλο του Κοινοβουλίου απλώς και μόνο στο σχολιασμό του ρόλου των, ε, του δικαστηρίου, αλλά του ε, δίνει στο δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να υποβάλει τις δικές του προτάσεις. Και εκτίμησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο εισηγητής δεν ε, αναφέρεται απλώς και μόνο στην απόρριψη ή στην αποδοχή των προτάσεων του δικαστηρίου, αλλά διατυπώνει και δικές μας προτάσεις, τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Τώρα, ας δούμε τα επιμέρους σημεία. Οι δύο πρώτες προτάσεις για την θέση του Αντιπροέδρου και της αύξησης των μελών της Ολομέλειας σε 15 είναι λογικές προτάσεις με τις οποίες είμαι σύμφωνος. Όμως θα ήθελα να ε, σχολιάσω λίγο τις άλλες δύο προτάσεις που υποβλήθηκαν. Καταρχάς όσον αφορά των προσωρινών δικαστών ή των αναπληρωτών δικαστών. Ε, συμφωνώ με τον εισηγητή, με τις απορίες που έχει ο εισηγητής δηλαδή, διότι και εγώ θεωρώ ότι καταρχάς θα πρέπει να έχουμε κατά νου το γεγονός ότι είναι δύσκολο να συγκρίνουμε στο σύνολό του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τους ε, οργανισμούς που το αποτελούν με το, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Και δεν μιλάμε για μια διεθνή συνθήκη, αλλά για ένα δικαστικό σύστημα ευρωπαϊκό. Επομένως όλες οι συγκρίσεις που γίνονται για αυτά τα θέματα θεωρώ ότι δεν είναι χρήσιμες. Να συγκρίνουμε δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και υπάρχει ένας κίνδυνος διαφοροποίησης του καθεστώτος που διέπει τους δικαστές. Εδώ μιλάμε για δικαστές ε, των ευρωπαϊκών κοινοτήτων που εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι δικαστή Οι δικαστές θα πρέπει να είναι όλοι το ίδιο. Επομένως αυτή η έννοια των προσωρινών ή αναπληρωτών δικαστών για το ε, Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης δεν με βρίσκει σύμφωνο. Επίσης, για το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Δεν ε, θεωρώ ότι, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έχει... Ε, δεν αμφισβητώ μάλλον το ότι έχει μια αυξανόμενη δουλειά, όμως εάν δείτε οι υποθέσεις που αντιμετωπίζει το δικαστήριο αυτό είναι κυρίως διπλώματα ευρωστεχνίας. Και τα διπλώματα ευρωστεχνίας δεν λύνονται, αν θέλετε, με μια αύξηση του αριθμού των δικαστών. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα που υπάρχει να δημιουργηθούν συγκεκριμένα δικαστήρια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να Δεν χρειάζεται να διευρύνουμε τι αρμοδιότητε του υπάρχοντο δικαστηρίου, ειδικού δικαστηρίου που είναι το Δικαστήριο Δημόσια Διοίκηση. Μιλήσαμε και προηγουμένως για την άμεση προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών εν γέννη. Που θα πρέπει να είναι δύο οι δικαστές, γιατί θα γίνουν 28 28, δικαστέ, 28 κρατημέλη, 28 δικαστές ε, θα πρέπει να γίνουν 30. Ε, θα πρέπει να, είναι και, να υπάρχει κάποιος παραπάνω. Ε, βέβαια δεν είναι οι δύο δικαστές, δεν είναι 12, αλλά τέλος πάντων. Το δικαστήριο θέλει να διατηρήσει τον ρόλο του ως εφετείο. Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, νομίζω ότι μπορεί, μάλλον ρυθμίζοντας κάπως τη λειτουργία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση του εισηγητή για τις απόψεις ε, της ε, μειονότητα, της μειοψηφίας, εγώ θεωρώ ούτως ή άλλως Υπάρχει αυτή η πρακτική στα δικαστήρια και συμφωνώ με τον εισηγητή στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά να σας πω ότι εγώ δεν ενθουσιάζομαι ιδιαίτερα με αυτή τη δυνατότητα, διότι εγώ θέλω ένα δικαστήριο όπου δεν θα υπάρχει μια υπερβολική πολιτικοποίηση των, του τρόπου λειτουργίας, ε, των αποφάσεων κτλ. και μπορεί η πρακτική αυτή να έχει τους λόγους της για το δηλαδή να ε, γνωστοποιείται η, απόφα... η γνώμη της ε, μειοψηφίας. Δηλαδή, καταλαβαίνω το πνεύμα με το οποίο έγινε η πρόταση του εισηγητή, αλλά έχω επιφυλάξεις. Και ολοκληρώνω διερωτώμενος μήπως ε, θα μπορούσαμε σαν ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσουμε τις αρμοδιότητές μας σαν, σαν, συναπο, σαν ε, όργανο της συναπόφασης αν θέλετε και να πούμε την άποψή μας για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εν γέννη. Υπάρχει και η θέμα της, το θέμα της εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ε, ακόμα εκεί δεν έχει δοθεί απάντηση. Επομένως, ίσως θα έπρεπε να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, ο κύριος Νταφ. Ναι, πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον συνάδελφο Μέσσερ Σμιτ για την για το σχέδιο γνωμοδότησής του. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το δικαστήριο αντιμετωπίζει μια μεγάλη αύξηση των ε, εργασιών του. Εν μέρη επειδή τρίφονται και κάποια θέματα πνευματικής διοκτησίας, εν μέρη επειδή ε, υπάρχει επέκταση του κοινωτικού της κοινωτικής νομοθεσίας στον τομέα των εσωτερικών ζητημάτων και των ζητημάτων δικαιοσύνης όπως είπε και ο κύριος Γκουατιέρη, αλλά και επειδή είναι επικείμενη προσχώρηση στην Ένωση Χάρτας Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο θα έχει συνέπειες και στο σύστημα του Λουξεμβούργου πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι το δικαστήριο θα έχει εξυγχρονιστεί επαρκώς προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ε, προσδοκίες μας σε ό,τι αφορά την ποιοτική και γρήγορη απόδοση δικαιοσύνης. Χρειάζεται λοιπόν μάλλον το Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να μην αποδεχτεί τις προτάσεις του δικαστηρίου, ιδιαίτερα όταν υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρέπει να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι προτάσεις του δικαστηρίου. Υπάρχουν φυσικά θέματα προϋπολογισμού. Αλλά φυσικά η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος έχει και κάποιο κόστος. Όπως και η δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά τους προσωρινούς ε, δικαστές, δεν συμφωνώ με την ανησυχία αυτή, ότι δηλαδή ακριβώς λόγω του προσωρινού χαρακτήρα τους είναι κατώτεροι. Πάντα γνωμοδοτείται σχετικά με την ε, ποιότητα των δικαστών. Πάντα υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ των δικαστών και γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δικαστές θα είναι μέλη, πρώην μέλη του δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά δηλαδή το τμήμα γενικών υποθέσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει βεβαιότητα σε σχέση με την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στο θέμα των επιπλέον δικαστών. Θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για την διαδικασία διορισμού. Είναι πολύ περίπλοκο ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά πρότεινε δύο λύσεις Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα τη δεύτερη λύση. Ξεκινώντας στην παράγραφο 49 της νομοδότησης, όπου κατανοείται φυσικά η ανάγκη εξειδικευσής προκειμένου να προκύψει ένα σύστημα διορισμού που θα επιτρέπει στους δικαστές να έχουν συγκεκριμένη εμπειρία και ειδίκευση σε κάποιον τομέα. Ο μόνος άλλος περιορισμός θα είναι ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα έχει πάνω από δύο δικαστές. Νομίζω ότι αυτό είναι εύλογο. Νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία εκπεριτροπής κατάληψη των θέσεων αυτών είναι λογική και νομίζω ότι θα πρέπει, αν συμφωνούμε με τη θέση αυτή, να το αναφέρουμε στη γνωμοδότηση. Σε περίπτωση αποκλίνοντων απόψεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαλεκτική μεταξύ των ε, των απόψεων των δικαστών και είναι δημόσια. Είναι δημόσιος ο διάλογος αυτός. Υπάρχει λοιπόν αυτό το στοιχείο της συζήτησης, της διαφάνειας. μιας διαδικασίας η οποία καταλήγει σε μια συνενετική άποψη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μια αποκλίνουσα άποψη θα αποσταθεροποιούσε την κατάσταση. Και την ε, ηρεμία των δικαστών στο Λουξεμβούργο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Τελευταίος. Α, δεν είναι τελευταίος. Ο κύριος Έφνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι να ευχαριστήσω τον κύριο Μέσσερ για την πολύ καλή δουλειά. Να προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω. Γιατί θα έχουμε άλλωστε και στο μέλλον ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά. Καταρχάς, υποστηρίζω την πρόταση για δημιουργία αξιώματος, θέσεις Αντιπρόεδρο και αύξηση του Γενικού Τμήματος από 13 σε 15 μέλη. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι μη αμφιλεγόμενο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μειοψηφικές ψήφους, σας υποστηρίζω. Θεωρώ ότι είναι καλή η πρότασή σας. Και όπως και ο κύριος ε, Γκουατιέρη, θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα αυτό του δικαστηρίου. Και θεωρώ ότι είναι σωστή η πρότασή σας. Δεν νομίζω ότι μειώνει αυτό το κύρος, την αξιοπρέπεια, την συνοχή της ατιμιγορίας. Γιατί έχουν νομική ισχύ οι δικαστικές αποφάσεις αυτές. Είναι θέμα διαφάνειας. Ωστόσο, συχνά έχουμε αποκλίνουσες ετοιμιγορίες από δικαστήρια, τα οποία, οι οποίες επηρεάζουν την ε, νομοθετική διαδικασία. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αποκλίνουσες απόψεις μπορεί να είναι πολύ καλά αιτιολογημένες και σε μετέπειτα χρονικό σημείο να επηρεάσουν την νομοθετική διαδικασία. Και ξέρω σε πολλές περιπτώσεις ε, ότι έχει εκφραστεί μια τέτοια αποκλίνουσα άποψη, η οποία έχει θεκτικό αντίκτυπο στο μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό μέσο και δεν νομίζω ότι δικαιολογείται το επιχείρημα της ε, ενιαίας ε, εικόνας του δικαστηρίου. Μία ερώτηση, μία παρατήρηση μάλλον να κάνω. Θα διατύπωνα με λίγο διαφορετικό τρόπο την αιτιολόγηση της θέσης αυτής, γιατί εδώ θέλουμε να καταλήξουμε σε μία γνωμοδότηση την οποία υποστηρίζει όλη η Επιτροπή. Νομίζω ότι στην αιτιολόγηση αυτά που αναφέρετε για την προσωπική σας άποψη σε ό,τι αφορά για θέματα ε, διακριτικής μεταχείρισης ήταν καλά. Αλλά γενικά θα ήθελα να μην συμπεριλαμβάνονται στο σημείο αυτό τέτοια προσωπικά παραδείγματα. Η ιδέα σας ωστόσο είναι σωστή, θεωρώ, για τον, την αύξηση των του αριθμού των δικαστών και σε ό,τι αφορά τη δημιουργία εξειδικευμένων τμήματων. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω ακόμα αποφανθεί, δεν έχω ακόμα αποφασίσει. Θα ήθελα καλέσω τον πρόεδρο, τον κύριο Καζίνη, να μας μιλήσει μήπως κι εσείς από την μακρά σας εμπειρία ως δικαστής μπορείτε να τοποθετηθείτε. Και τέλος μία ερώτηση στον Μόρτεν Μέσσερ Σμιτ, το ανέφερε και ο κύριος Ντάφ, σε ό,τι αφορά το θέμα της, του διορισμού. Γιατί δεν τοποθετηθήκατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγγελ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάρτιν για το σχέδιο γνωμοδότησης. Κατά την άποψή μου είναι καλό και συνεκτικό. Έχω άποψη για κάθε ένα από τα θέματα που συζητήσαμε εδώ, αλλά θα περιοριστώ σε δύο πράγματα. Το ένα είναι το θέμα της διεύρυνσης της σύνθεσης του δικαστηρίου δεν είμαι κατά της αύξησης του αριθμού των δικαστών ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά θεωρώ ότι καλό είναι να υπάρχει ένα δικαστήριο το οποίο να μην έχει πολύ μεγάλη σύνθεση. Αν θέλουμε να έχουμε ειδικά δικαστήρια διαφορετικών μορφών για να αντιμετωπίσουμε το φόρτο εργασίας και τις υποθέσεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, καλός. Αλλά πρέπει να έχουμε ένα περιορισμένο δικαστήριο. Δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη σύνθεση του δικαστηρίου και πρέπει να ε, αφορά τα βασικά ζητήματα. Αν θέλουμε να ξανασκεφτούμε τον αριθμό των δικαστών, θα πρέπει ίσως να δούμε και πιο θα πρέπει να είναι το ανώτατο όργανο του δικαστικού συστήματός μας. Δεύτερον, υποστηρίζω πλήρως την ιδέα της αποκλίνουσας γνώμης και της ε, κοινοποίησης ε, των αιτιάσεων κάθε δικαστή ή τέλος πάντων όποιου δικαστή θέλει να αποκαλύψει την άποψή του. Αναφερόμαστε συνεχώς στη δημοκρατία και στη νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα προβλήματα της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο κρατών μελών είναι η νομιμότητα του δικαστικού συστήματος. Όχι σε όλες τις χώρες, αλλά σε μεγάλο αριθμό χωρών είναι πρόβλημα και θεωρώ ότι επειδή ακριβώς αυξάνεται η σημασία του δικαστικού συστήματος στην κοινωνία μας, θα αποτελέσει και μείζον θέμα στις ευρωπαϊκές χώρες. Οτιδήποτε λοιπόν μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να ενισχύσουμε την νομιμότητα και το δημοκρατικό χαρακτήρα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του δικαστηρίου είναι καλώς καμωμένο. Υποστηρίζω πλήρως λοιπόν το θέμα αυτό και με το επιχειρήμα της δημοκρατικής νομιμότητας. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει να παρουσιάζονται όλες οι απόψεις, όλες οι γνώμες, όλα τα επιχειρήματα και τότε η απόφαση αυτή μπορεί να γίνει αποδεχθεί ευρύτερα. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε άλλωστε ότι ότι στο ευρωπαϊκό νομικό σύστημα έχουμε νομολογία. Βασιζόμαστε στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Επομένως, η δημοκρατική νομιμότητα του δικαστηρίου είναι πολύ πιο σημαντική από ε, ένα σύστημα όπου έχουμε common law, έχουμε Τα θέματα λοιπόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι κατά βάση νομολογία δικαστηρίου. Δεν είναι ένα σύστημα ε, αστικού δικαίου. Γι' αυτό λοιπόν τα πάντα βασιζόμαστε στις δικαστικές αποφάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αυξηθεί η νομιμότητα του δικαστηρίου και να δεχτούμε το θέμα της αποκλίνουσας γνώμης. Γιατί αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας του δικαστηρίου. Έχω Ωραία. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μέσσερ Σμιτ να απαντήσει, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την άποψή μου για το θέμα των αντιπροέδρων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι καλό ήταν να υπάρχει ένας αντιπρόεδρος που να μπορεί να αντικαθιστά τον πρόεδρο. Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Τώρα, για το θέμα των ε, προσωρινών ε, δικαστών. Εγώ δεν θεωρώ ότι μειώνεται το βάρος του δικαστηρίου εάν υπάρχει κάποιος αναπληρωτής δικαστής σε όλα τα νομικά, τα δικαστικά συστήματα, αν θέλετε, μπορούν να, στην Ιταλία τουλάχιστον, μπορούν να λειτουργήσουν ε, δικαστές που ε, δεν είχαν οριστεί από την αρχή. Αρχή, βέβαια να, ορί, να διορίζονται με έναν ε, σωστό τρόπο. Ούτως ή άλλως το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το δικαστικό σύστημα στην Ευρώπη είναι η βραδύτητα μία απόφαση του δικαστηρίου, ενός δικαστηρίου, είναι να έχουμε σωστές αποφάσεις. Δηλαδή να έχουμε μέγιστες εγγύσεις για να έχουμε σωστές αποφάσεις. Το πρόβλημα είναι η βραδύτητα. Άρα, εάν μπορούμε να έχουμε μέγιστες εγγύησεις όσον αφορά το σωστό της, ε, της σύνθεσης και να λειτουργεί γρήγορα το δικαστήριο, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι οι εγγύσεις σε διορισμό αυτών των ε, δικαστών. Τώρα, υπάρχει και θέμα ε, ισορροπίας των συμφερόντων. Υπάρχει ένα... Υπάρχει με ένα πολιτιστικό θέμα, αλλά πιστεύω ότι αυτόν τον, το θέμα των προσωρινών δικαστών είναι το, μπορεί να τεθεί μόνο σε περίπτωση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. Το, συγγνώμη, ε, η, η, άποψη της μειοψηφία είναι και θέμα ε, πολιτιστικό, αν θέλετε. Κάθε χώρα έχει τη δική της κουλτούρα. Αλλά εγώ προτιμώ την ανωνυμία, αν θέλετε. Την ανωνυμία των δικαστών. Δηλαδή, σε θέματα δικαιοσύνης είναι το όργανο το οποίο μετράει, όχι το άτομο. Στην Ιταλία έχει γίνει η προσωποποίηση των δικαστών, υπερβολική προσωποποίηση και αυτό είναι επικίνδυνο, διότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να επηρεαστεί και η ανεξαρτησία του δικαστή. δεν ξέρει πώ μπορεί να αντιδράσει όταν υπάρχουν απειλέ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι από, διάφορους, από διάφορους κύκλους. Επομένως, καλό θα είναι ο δικαστής όταν δικάζει να έχει όλες τις εγγυήσεις ότι μπορεί να ε, πάρει την απόφασή του ανεξάρτητα. έχοντας την μέγιστη δυνατή εγγύηση ανεξαρτησίας. Και βλέπω τι γίνεται στην ε, Ιταλία και με τις διάφορες εισαγγελίε, ας πούμε. Όταν μιλάμε, όταν γίνεται μια έρευνα, είναι η εισαγγελία της Ρώμης, όχι ο εισαγγελέα. Είναι η εισαγγελία, είναι το όργανο δηλαδή. Γιατί τα άτομα μπορεί να είναι τα άτομα μπορεί να είναι δεξιά, αριστερά, κεντρό, να έχουν άλλες αποχρώσεις κτλ. Ενώ το όργανο αποφασίζει. Μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε. Δεν μπορούμε να λέμε το Ευρωπαϊκό ε, Δικαστήριο αποφάσισε, αλλά ο Αυστριακός δικαστής είπε αυτό. Ο Κροατίς δικαστής είπε το άλλο. Ο Κροάτη. ο είπε το, το, το άλλο. Δεν, δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειε. Το δικαστήριο αποφασίζει. Και ελπίζω και ότι ο Γκολτιέρη να συμφωνεί. Τώρα να τα και από τα συστήματα, διότι υπάρχουν ε, νομικά, δικαστικά συστήματα όπου η άποψη της μειοψηφία είναι ε, θεσμός. Εγώ όμως προτιμώ να αποκλειστεί το οποιοδήποτε ενδεχόμενο επιρροής πάνω στους δικαστές, διότι πιστεύω ότι πραγματικά ε, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο και η απόφαση. Τώρα, θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τον συνάδελφο μέσα σου να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και για τα επικοδομητικά σας σχόλια. Κύριε Γκολιθιέρη, βλέπω ότι από τις περισσότερες προτάσεις από το δικαστήριο συμφωνούμε, όμως φαίνεται ότι εσείς προτιμάτε το σύστημα των ειδικών δικαστηριών. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο το προτιμάτε, αλλά κατά την άποψή μου δεν θα βοηθήσει το φόρτο εργασίας του δικαστηρίου διότι θα χρειαστεί πολλής χρόνος για να συσταθούν αυτά τα νέα ειδικά δικαστήρια και μπορεί σε τρία-τέσσερα χρόνια ή όταν τέλος πάντων ρυθμιστεί το, το ζήτημα θα αρχίσει τότε να μειώνεται το, το άφθος εργασίας, αλλά το πρόβλημα υπάρχει ήδη τώρα, επομένως πρέπει να βρούμε μια λύση για το παρόν. Ίσως θα ήταν καλό να ανοιχτεί αυτό ως ενδεχόμενο για το μέλλον, αλλά να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα προς το παρόν. Είμαι ε, ανοιχτό σε προτάσεις στην αναθεώρηση του κειμένου μου. Για τις άλλες προτάσεις, το, προτάσεις σας τώρα θα δω εάν πρέπει να τις συμπεριλάβουμε και αυτές. Τώρα, για το θέμα της αποκλίνουσας γνώμης. δεν ε, ε, καταλαβαίνω ότι το βλέπετε ως πλήρες βέτο. Κατάλαβα ότι διστάζετε για την ιδέα αυτή. Ε, και υπάρχουν διαφορές βεβαίως ε, μεταξύ του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, πρέπει να τηρούνται οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Είναι πολύ πιο επίσημα τα όσα έχουμε σε σχέση με το Στρασβούργο. Ε, εν τέλει όμως θεωρώ ότι Πολλές από τις ε, υποθέσεις ε, όσον αφορά την εργόρα εργασίας, για παράδειγμα, τις διακρίσεις, συμφωνώ ε, ότι τα δύο αυτά θέματα αντιμετωπίζονται και από τα δύο δικαστήρια. Ως πολιτικός, αλλά και ως νομικός, νομίζω ότι έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της πρόθεσης του δικαστηρίου, αν υπάρχει δυνατότητα να εξηγήσουν επακριβώς πού υπήρχε η διαφωνία στο δικαστήριο στις συζητήσεις μεταξύ δικαστών. Όλοι γνωρίζουν ότι οι δικαστές, όπως και οι πολιτικοί, όπως και οποιοδήποτε άλλος, ε, διαφωνούν. Ε, σε τεχνικά ζητήματα ορισμένες φορές. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν πολλές αποφάσεις που αποτελούν ε, συμβιβασμό και δεν είναι σαφές ε, τι ακριβώς ε, θέλαμε στην απόφαση και το πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό. Εάν υπάρχει λοιπόν μία μικρή μειοψηφία ή ένας-δύο δικαστές που μπορεί να πούν ότι διαφωνούν με την πλειοψηφία, αλλά θεωρούν ότι αυτό θα έπρεπε να ισχύει και επομένω όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να γνωρίζουν επακριβώς ποια είναι η άποψη του δικαστηρίου. Και αυτό ακριβώ γίνεται στο Στρασβούργο. Και Αυτό οδήγησε σε μια σαφέστερη θέση για την πρόθεση του δικαστηρίου και γι' αυτό ακριβώ έκανα την πρόταση αυτή. Θα μπορούσα να αναφερθώ και στα πολλά κράτη-μέλη που έχουν το σύστημα αυτό. Ε, ξέρω ότι η Ιταλία δεν διαθέτει ένα αντίστοιχο σύστημα, αλλά πολλέ άλλε χώρε το διαθέτουν. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία, ε, και αυτό ακριβώ πρότεινα εδώ στο σχέδιο γνωμοδότηση είναι να μην είναι υποχρεωτικό, απλώς να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν οι δικαστές. Όπως σας είπα όμως, δεν θεωρώ ότι αγνοείται πλήρως την ιδέα, ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσετε. Ο κύριος Νταφ τώρα. Μπορεί να έχει δίκιο ότι ε, το κοινοβούλιο μπορεί να απορρίψει και απόψεις του δικαστηρίου, τις οποίες υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θεωρώ ότι καλό είναι να σκεφτούμε τουλάχιστον ε, στη γνωμοδότηση κάποιες από τις ανησυχίες που εξέφρασε το δικαστήριο. Δεν είναι απαραίτητο να δεχτούμε ή μάλλον να το θέσω αλλιώς. Μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση του δικαστηρίου εκφράζοντας και την ανησυχία μας για το πού μπορεί να οδηγήσει ε, το θέμα των ε, αναπληρωτών δικαστών, επί παραδείγματι. Επειδή σας είπα και επεσήμενα ποιο είναι το πνεύμα της συνθήκης κατά την άποψή μου όσον αφορά τη διαφάνεια, με εκπλήσει το γεγονός ότι ο κύριος Ντάφ είναι κατά της άποψης της αποκλίνουσας γνώμης και να έχουμε μόνο την ε, έκδοση της απόφασης της πλειοψηφίας. Ορισμένες φορές ε, ε, μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τον Γενικό Εισαγγελέα, αλλά ο Εισαγγελέας δεν έχει κάποια εντολή όπως έχουν οι δικαστές και δεν είναι σαφές εάν οι δύο αυτές θέσεις αντικατοπτρίζουν όλες τις συζητήσεις που έγιναν εντός του δικαστηρίου. Μπορεί πολύ εύκολα να υπάρχει ένας μειοψηφικό αριθμό δικαστών που να είναι της άποψης ότι δεν ε, εκφράζει η άποψή τους από αυτό που λέει ο Γενικός Εισαγγελέας παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει διαφωνία μεταξύ της πλειοψηφίας του δικαστηρίου και του εισαγγελέα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί το δικαστήριο να ακολουθήσει την άποψη του εισαγγελέα, αλλά να υπάρχει μια ομοιοψηφική θέση δικαστών που να έχει διαφορετική άποψη για την ερμηνεία του κεκτημένου και να μην τους δοθεί δυνατότητα να εισακουστούν. Και αυτό βέβαια από πλευράς ε, διαφάνειας και πιο ανοιχτής άποψης μπορεί να δημιουργεί θέμα και εκτιμένου, γιατί μπορεί να είναι μια μειοψηφία η οποία πρέπει να βρει έναν τρόπο να συμφωνήσει με την πλειοψηφία ε, και αυτό φυσικά δημιουργεί πρόβλημα και για την πλειοψηφία που είναι υπέρ μια άποψη, γιατί πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συμβιβαστούν. Ευχαριστώ τον κύριο Χέφνερ για την υποστήριξή του για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα το πώς ε, διορίζονται οι δικαστές, ε, το σημειώνω, θα βρω έναν τρόπο να το δούμε αυτό και άλλοι έχουν εξετάσει το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να δούμε τη διαδικασία για να ε, διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις εγγυήσεις που ανέφερε και ο πρόεδρος στην παρέμβασή του. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει φυσικά και για τους αναπληρωματές δικαστές και θα το αναφέρω αυτό στο κείμενό Να ευχαριστήσω και τον κύριο Ράνκελ για τα σχόλιά του και την υποστήριξή του για την ε, ε γνωμοδότησή μου και τη σαφή ανάλυση της ιδιαιτερότητας του δικαστικού συστήματος που είναι ένα σύστημα ε, νομολογίας για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτό φυσικά μας δίνει τη δυνατότητα οι δικαστές να είναι σαφείς για το ποια είναι η άποψή τους ε, για ένα θέμα. Και τέλος, ως απάντηση στα όσα είπε ο Πρόεδρος, κατανοώ την άποψή σας ότι το όργανο είναι αυτό το οποίο εκφράζει την απόφασή του, επομένω θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία των δικαστηρίων, αλλά ορισμένες φορές με τη σύνθεση που έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πολλές φορές οι αποφάσεις οι οποίες εκδίδει είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και θα ήταν δίκαιο να είναι ε, πλήρης η διαφάνεια για τις συζητήσεις που διεμήφθησαν πριν από την έκδοση μιας απόφασης. η ανωνυμία δεν διασφαλίζει απαραίτητα την πλήρη ανεξαρτησία. Τα μέλη του δικαστηρίου ούτως ή άλλως πρέπει να ορίζονται από τα κράτη-μέλη και δεν ε, βλέπω πώς η ανωνυμία διασφαλίζει την ανεξαρτησία επειδή δεν υπάρχουν αποκλίνουσες γνώμες. Ξέρω πολύ καλά ότι ως δικαστής ε, έχετε μακρά πείρα και θα πρέπει να βασιζόμαστε και στην δυνατότητα που έχει ο δικαστής να προασπίσει και το δικαστήριο, αλλά και να ερμηνεύει ορθά την νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε ότι οι δικαστές ε, οι οποίοι είναι αυτοί αποφασίζουν για το πώς ερμηνεύεται το κοινοτικό κεκτημένο έχουν την ανάγκη να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία. Νομίζω ότι οι δικαστές που διαδραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο και δικαίως για το θέμα αυτό, ε, θα πρέπει να δίνουν στο δικαίωμα στο κοινό να έχει πλήρη πρόσβαση ε, για την έκδοση μιας απόφασης. Αυτό δεν ε, μειώνει τη βαρύτητα οποιοδήποτε δικαστηρίου ε, χώρας μέλος που έχει αυτό το σύστημα, ούτε μειώνει τη βαρύτητα του δικαστηρίου στο Στρασβούργο, ε, και σε καμία περίπτωση δεν θα μειώσει τη βαρύτητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ίσα ίσα θα του δώσουμε λιγότερη νομιμότητα, λιγότερη διαφάνεια από όσοι μπορεί να βρει οποιοδήποτε πολίτη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Ε, έχουμε αποφάσει σε ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο θα υπερβαίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τουλάχιστον εξ όσων αντιλαμβάνομαι εγώ την παρούσα συμφωνία. Επομένως, νομίζω ότι θα είμαστε σε δύσκολη θέση εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μπορεί να δώσει τις ίδιες εγγύησεις διαφάνειας που ε, διαπιστώνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Ε, άκουσα τα όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι, θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο κειμένου και φυσικά ε, περιμένω να κάνουμε και περιττέρω συζητήσεις επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μέσσερ Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα πρέπει να ορίσουμε την ημερομηνία για την υποβολή των ε, τροπολογιών. Πιστεύω Τι είχαμε προβλέψει, 27 Οκτωβρίου. Λοιπόν, ψηφίζουμε 22 Νοεμβρίου, άρα την ε, προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 27 Οκτωβρίου. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μας. Να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 24 ε, Οκτωβρίου. Είναι, θα είναι στο Στρασβούργο, είναι έκτακτη 21 ε, Νοεμβρίου, έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.